Hello to everybody. Good morning. Καλημέρα σε όλους σας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά το διάλειμμα που φαίνεται τόσο μακριά και δεν έγινε ποτέ. Καλή χρονιά φυσικά. Ε, έχουμε αργήσει λίγο, φτάνουμε τέλη Ιανουαρίου, αλλά προλαβαίνουμε ακόμα να λέμε τα χρόνια πολλά. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε προτάσεις, τίποτα. Ε, ο κύριος Πάτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλή σας χρονιά σε όλους. Έχω μια ερώτηση στην ημερήσια διάταξη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε προβλέψει κάποιο χρόνο για την επιστολή σας σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ έχω εδώ την επιστολή που λέγει ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέτασε το θέμα στις 22 Ιανουαρίου του 2020. Σήμερα είναι αυτό. Και κοίταξα την ημερήσια διάταξη είδα τις ψηφοφορίες, αλλά δεν είδα να έχετε προβλέψει χρόνο για εξέταση, συζήτηση, τίποτα. Αυτή η γνωμοδότηση υπομορφή επιστολής είναι γνωστή εδώ και πέντε μήνες, γιατί τότε λήφθη η απόφαση από τους συντονιστές ότι θα απαντήσουμε στο αίτημα για γνωμοδότηση και επί πέντε μήνες έχουμε συνεδριάσεις και συνεδριάσεις εκτός της Επιτροπής με εισηγητές και τα λοιπά και μόλις προχθές είδαμε το σχέδιο το τελικό. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να κάνω ούτε τροπολογία ως μη εγγεγραμμένος, ούτε να συμμετάσχω σε διάφορες συζητήσεις και η Επιτροπή μας ποτέ δεν το εξέταξε αυτό. Και στην ημερήσια διάταξη βλέπω ότι συζητάμε διάφορα πράγματα. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλά στο παρελθόν. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τουλάχιστον τρεις φορές, δύο φορές το έχουμε συζητήσει, έτσι και αλλιώ, ε, για τα διπλώματα οδήγηση και τον ΚΟΚ και τα λοιπά. Νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό θα ε, παρακαλούσα να τα χρόνο στην ημέρησα διάταξη πριν την ψηφοφορία που μπορεί να μετατεθεί για να συζητήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση Παύλα επιστολή σας. Ευχαριστώ. Any remarks from the... Άλλα σχόλια από τους συντονιστές για αυτό το θέμα. It's so ε, όχι. Ωραία, σημειώνουμε το σχόλιο σας, κύριε ε, Πάτεν. Κατανοώ τα όσα λέτε. Διαδικαστικά μόνο να σας πω το εξής. Η διαδικασία αυτή καθ' αυτή ήταν απόλυτα διαφανής, καθώς είστε ενήμερος κι εσείς. Ενδεχομένως, αν έχετε ενδιαφέρον, να το συζητήσουμε το απόγευμα που συνεδριάζουν οι συντονιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, με κάθε σεβασμό, τι μας λέτε τώρα. Πριν τις ψηφοφορίες υπάρχει καμία περίπτωση να το συζητήσουμε ή θέλετε μετά τις ψηφοφορίες. Η κυρία Ραφάλσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι αυτό το θέμα ε, χρειάζεται να το δούμε σε βάθος. Αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να το συζητήσουμε και δεν επηρεάζει πολύ την ημερήσια διάταξη, θα παρακαλούσα να αλλάξει η ημερήσια διάταξη, να πάρουμε σοβαρά αυτή την πρόταση και να τη δεχτούμε, να το συζητήσουμε το θέμα. Yeah, unfortunately... Δυστυχώς, αυτό το θέμα μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά μόνο μετά την ψηφοφορία, όχι πριν την ψηφοφορία. Τι να κάνουμε τώρα, το ξέρω ε, πώς ακούγεται αυτό. Έχω απόλυτη επίγνωση, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν χωράει άλλη συζήτηση για αυτό το θέμα χρονικά πριν τις ψηφοφορίες της σημερινής συνεδρίαση. Ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Κροατική Προεδρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καλωσορίζω λοιπόν σήμερα τους ε, δύο υπουργούς, τον κύριο Γιώσιπ Αλαντρόβιτς, ε, Υπουργό Εργασίας και Συντάξεων, και την κυρία Βέσνα Μπεντέκοβιτ, Υπουργό Δημογραφία, Οικογένεια, Νεολαία και Κοινωνικής πολιτική. Θα μας παρουσιάσουν σήμερα το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας. Γνωρίζουμε πως ε, η Προεδρία αντιμετωπίζει πολλές ε, προκλήσεις μεταξύ των οποίων το Brexit, τον προϋπολογισμό 2021-2027, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε και κάποιους ε, νομοθετικούς ε, φακέλους που δεν έχουν κλείσει. Το ένα και μοναδικό συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ε, που θα σας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει και σήμερα θα θέλαμε να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα για τις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας που νομίζω ότι ταυτίζονται με τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν. Δίνω τον λόγο στον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που βρισκόμαι σήμερα εδώ μαζί σας ε, για να παρουσιάσω τις ε, πολιτικές μας μαζί με τον Πρωθυπουργό Μπεντεκοβιτς στο Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι η πρώτη μας Προεδρία και είμαστε ιδιαίτερος υπερήφανοι για το ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τα όσα θέλουν οι πολίτες μας από εμάς, δηλαδή ποιότητα ε, θέσεων εργασίας, αξιοπρεπής μισθή σε κάθε μέρος της Ευρώπης. Για την Κροατία, το νεότερο κράτος μέλος, έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε νέες εμπειρίες και να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Πριν παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας, θα ε, δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω την Ρουμανική και Φιλανδική Προεδρία για όλες τις ε, προσπάθειές τους. Το πρόγραμμα της ε, Κροατικής Προεδρίας βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες, τα κοινά συμφέροντα και τον σεβασμό της διαφορετικής άποψης. Στο επίκεντρο είναι οι ανάγκες των πολιτών μας για ασφαλεία και ποιότητα ζωής. Γι' αυτό ακριβώς κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας ε, θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε πρόοδο στα ζητήματα αυτά τα οποία επηρεάζουν ε, τις συνθήκες εργασίας και τις ζωές των πολιτών μας. Η Κροατία έχει τέσσερις κύριες προτεραιότητες. με Ευρώπη που συνδέει, που προστατεύει, που ασκεί επιρροή και που αναπτύσσει. Και αναπτύσσεται. Οι προτεραιότητες μας είναι αναπτυξιακές προτεραιότητες γιατί χωρίς ισχυρότερη σύγκληση και μια μεγαλύτερη ανάπτυξη δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο για τις επόμενες γενιές. Για τον λόγο αυτόν είμαστε πεπισμένοι ότι η περαιτέρω εφαρμογή του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι μια καλή βάση για τις ε, μελλοντικές μας ε, προσπάθειες και η Κροατική Προεδρία θα προσπαθήσει να πετύχει μια ευρεία εφαρμογή των αρχών αυτών. Και είμαστε πεπισμένοι ότι θα μας στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ακριβώς το θέμα της κοινωνικής συνοχής ως βασικό παράγοντα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών μας. Η ευημερία της Ένωσης ακόμα δεν ε, έχει διαχυθεί ομοιόμορφα προς όλους και θα πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε τρόπους να συμβεί αυτό και να φροντίσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή για να έχουν καλύτερες προοπτικές ε, ένταξης ε, και στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας της Ένωσης αντιμετωπίζει έλλειψη δικευμένων εργαζομένων και πρέπει να επιληθεί αυτό για να έχουμε ανταγωνιστικότητα παγκοσμίω. Οπότε η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αναπτυξή των δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα, για την ανταγωνιστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, συνολικές ανάγκες για τον 21ο αιώνα. Πρέπει ακριβώς ε, να παρακολουθούμε στην ευρωπαϊκή οικονομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις ε, παράλληλα με τις άλλες μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Οι ψηφιακές δεξιότητες, η κριτική ικανότητα, η ικανότητα επίλυσης ε, προβλημάτων είναι πράγματα που απαιτούνται πλέον από το εργατικό δυναμικό. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσει η συζήτηση για το πώς θα ταιριάσουν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας ε, με την διαβίου εκπαίδευση εργαζομένων και μη. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να βρεθούν βιώσιμοι τρόποι χρηματοδότησης, γιατί η ψηφιοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί συνεχή ενημέρωση των δεξιοτήτων. Γι' αυτό προτείνουμε να έχουμε και κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα των δεξιοτήτων και μαζί με αυτό θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα σε μια υπουργική διάσκεψη στις 12 και 13 Μαΐου στο Ντουμπρόβνικ. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τα μελλοντικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και για τον λόγο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ. Παρά το ότι η Ευρώπη έχει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας στον κόσμο, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. επίσης για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, ε, στην τεχνολογική πρόοδο και τις νέες μορφές εργασίας πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Υπάρχουν διάφορες πτυχές ε, καινοτόμων μορφών εργασίας και πρέπει βεβαίως να συζητήσουμε με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Η εξέβρεση λύσεων είναι σημαντική για όλα τα κρατημέλη. στόχο είναι να διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε ποιοτικέ θέσει εργασία και να αυξηθεί η προστασία των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνεται η ισορροπία ιδιωτικού και εργασιακού βίου. Αυτά βεβαίως σκοπεύουμε να τα συζητήσουμε για να μπουν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Σκοπεύουμε λοιπόν να κάνουμε διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οικονομία και την κοινωνική διάσταση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους μας και είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι απόψεις. Για να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη και ένα καλύτερο μέλλον, οι πολιτικές μας πρέπει να προκύπτουν από διάλογο, συμφωνία και τήρηση των κανόνων. Για να υλοποιήσουμε τους κοινούς μας στόχους σε ένα πνεύμα συνεργασίας και φιλίας για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να είμαστε ισχυροί σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να δώσω τώρα τον λόγο στην ε, κυρία Υπουργό, την κυρία Μπεσακοβίτση. Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Νικότσοβα. Κυρίε και κύριοι, συντονιστέ των πολιτικών ομάδων, Είναι μεγάλη τιμή για μένα και ταυτόχρονα μεγάλη ευχαρίστησή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί με τον συνάδελφο Υπουργό Εργασίας Όπως γνωρίζετε μετά από 6,5 χρόνια, μετά την ένταξη της χώρας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήραμε πλέον τη σκητάλη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μου. θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τα πιο βασικά στοιχεία των δραστηριοτήτων τις οποίες προβλέπουμε να αναλάβουμε τους επόμενους μήνες στον κοινωνικό τομέα. Θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στους τομείς στους οποίους με στρατηγικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει προστιθέμενη αξία δημιουργώντας μια αίσθηση ισότητας στους πολίτες της, αλλά και ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα κοινών αρχών στα πλαίσια του νέου πλέον θεσμικού και νομοθετικού κύκλου στον οποίο μπαίνουμε. Έχουν ανανεωθεί και οι εντολές του Συμβουλίου και ε, οι θέσεις φυσικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπαίνουμε σε μια νέα φάση χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο και μπορούμε να συγκρίνουμε νομίζω και να συζητήσουμε τις προτεραιότητές μας για τα επόμενα χρόνια. Η Κροατία έχει ήδη προετοιμάσει το πρόγραμμά της σε τέσσερις πυλώνες τους οποίους προανέφερε ο κύριος Αλάντροβιτς. Κατά τη διάρκεια του επομένου εξαμήνου λοιπόν θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας πριν από οτιδήποτε άλλο στην προσπάθεια ενίσχυσης της Ευρώπης. Αυτός είναι και ο στόχος μας, αυτό είναι και το σύνθημά μας. Αποκινούμε τον συνάδελφο Αλάντροβιτς θα συμπροεδρεύσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών ΕΠΣΚΟ για να ακούσουμε και τις προτεραιότητες των μεμονωμένων κρατών μελών. Δύο είναι οι βασικές προτεραιότητες μας. Καταρχάς, το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής και η δημογραφική πρόκληση. Το άλλο θέμα είναι πάντα η ισότητα ανδρών και γυναικών και η βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σε σχέση με το δημογραφικό θέμα, τη δημογραφική πρόκληση καλύτερα, η κοινωνική πολιτική χαρακτηρίζεται θα έλεγα από το ότι τα περισσότερα από, μισά, από τα μισά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν θέματα δημογραφικά αρκετά δύσκολα και αυτό ε, φαίνεται και στο στρατηγικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2024. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε τις πολιτικές μέσω των οποίων θα είναι δυνατόν να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε τις οικογένειες και να βοηθήσουμε τις οικογένειες να συνδυάσουν καλύτερα την επαγγελματική ζωή, την επαγγελματική δραστηριότητα με την οικογενειακή διαχείριση. Αυτά είναι θέματα ε, τα οποία εν πωλής εξαρτώνται και από τα κράτη-μέλη και εξαρτάται από τις αρμοδιότητες τις οποίες έχουν τα κράτη-μέλη. Τι μπορούμε λοιπόν από κοινού να κάνουμε εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πολιτικές μπορούμε να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την λειτουργία, την εύρυθμη των κοινωνικών υπηρεσιών προς όφελος και εξυπηρέτηση των οικογένειών. Θυμίζω ότι δυστυχώς τα περισσότερα από τα φαινόμενα τα οποία είναι συνέπεια των δημογραφικών προβλημάτων θίγουν κυρίως τους ε, λιγότερο ισχυρούς οικονομικά. Όπως είπα η δεύτερη προτεραιότητά μας είναι οι γυναίκες και η αγορά εργασίας. Η καλύτερη ε, παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι προϋπόθεση για την αυτονόμηση των γυναικών και για την βελτίωση της θέσης τους κοινωνικά και γενικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και την οικονομική ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν να αυξήσουμε το ποσοστό των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε κατά κάποιο τρόπο ε, τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν ε, οι γυναίκες με το μεγάλο ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται εκτός εργασίας. Τίθεται το θέμα της εξάρτησης επίσης ε, μιας κατηγορίας πολιτών, γυναικών από τα συστήματα προστασίας τα οποία κανονικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα. οι κοινωνικές υπηρεσίες και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες επηρεάζουν εν πολλής τη ζωή των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να βελτιώσουμε την παροχή αυτών των υπηρεσιών και φυσικά να βελτιώσουμε και την παρουσία των γυναικών στον, στην αγορά εργασίας να καλύψουμε τη διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών και να προωθήσουμε επίσης και άλλους παράγοντες οι οποίες θα διευκολύνουν την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Θα οργανώσουμε επίσης και μια υπουργική διάσκεψη για τις δημογραφικές προκλήσεις και τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 Απριλίου 6 και 7 Απριλίου θέλουμε να δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε να γίνει επιτέλους μια ισχυρή, μια σοβαρή έντονη συζήτηση για τις δημογραφικές τάσεις στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να προτείνουμε και πιθανές λύσεις σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετά από τα, από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, για την αναπηρία 8 με 10 Μαΐου θα κάνουμε μία διάσκεψη όπου θα συζητήσουμε εκ νέου τα θέματα των δικαιωμάτων των αναπήρων. Μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις είναι αυτή η οποία θα θέσει το θέμα της ε, ε, κατάσταση, συνολικά της κατάστασης της παιδικής ηλικία και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η παιδική ηλικία, των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Και θα προσπαθήσουμε να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές στις χώρες μας. Στα πλαίσια του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ, ανεπίσημα, στις 26 και 27 Απριλίου, θα θέσουμε επίσης ε, θέματα που άπτονται τις σχέσεις απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Ήταν κάπως σχηματικά ε, τα πρώτα στοιχεία, αν θέλετε, ε, της δράσης την οποία σκοπεύουμε να αναλάβουμε τους επόμενους μήνες. Να υπογραμμίσω επίσης ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με υψηλές ταχύτητες. συνειδητοποιούμε απόλυτα τις προκλήσεις τις οποίες δημιουργεί η σύγχρονη κοινωνία και θέλουμε να λειτουργήσουμε σαν αντικειμενικός διαμεσολαβητής και γι' αυτό θα κάνουμε κάθε προσπάθεια η οποία θα έχει σαν στόχο την βελτίωση του επίπεδου ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαι βεβαία ότι θα συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας για τις σύντομες παρουσιάσεις της κρατικής προεδρίας. Ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων θα γίνει τώρα από τους συντονιστές και πρώτος γύρος απαντήσεων και μετά τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα ρωτήσουν και θα απαντηθούν οι ερωτήσεις. Ο κύριος Ράτκε πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Αναλαμβάνετε τη σκητάλη, παραλαμβάνετε τη σκητάλη. Μήπως να περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας. It, works now. Ακούτε τώρα. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι αναλαμβάνετε τώρα την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια δύσκολη περίοδο και κατάσταση. Έχετε πολλά πράγματα να ε, διεκπαιρεώσετε. Αναφερθήκατε σε αυτά. Θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το γεγονός ότι αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το παρουσιάσατε ως επιτυχία. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω ε, πώς βλέπετε τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε ε, διάφορες φήμες που κυκλοφορούν ότι θα πάρουν πόρους από εκεί για να πάνε στο ε, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το νέο που συστήνεται. Εγώ καλωσορίζω φυσικά την ίδρυση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, αλλά δεν θα παίρνουμε από την αριστερή τσέπη να τα βάζουμε στη δεξιά με διάφορες μεταφορές πιστώσεων με έναν έτσι αυτοματισμό ε, μίας ενδιαφερόμενης ομάδας απέναντι στην άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα. Αυτό το αποκρούω και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας θέση και πώς βλέπετε τις εξελίξεις της διαπραγματεύσεις. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ε, κάτι άλλο που αναφέρατε είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Μάλιστα πολλές φορές ε, το τονίσατε και το αναγνωρίσατε και σας ευχαριστώ γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κοινωνικούς εταίρους ισχυρούς και σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης για να μπορούν να λύνονται πολύ κομβικά προβλήματα, ε, ιδιαίτερα ε, μισθολογικού χαρακτήρα. Τι λέει λοιπόν η Κροατική Προεδρία για το θέμα του Ευρωπαϊκού Κατώτατου Μισθού. Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να έρθει ε, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας εκεί θα είναι επίκαιρη ας πούμε, αλλά οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους έχουν ήδη ξεκινήσει. Ε, είναι της δικής σας αρμοδιότητας, οπότε θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μάθω ε, ποια είναι η θέση της Κροατικής Προεδρίας. Και αν προωθείτε το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι πρόθεσή σας αυτό. Και μια συγκεκριμένη ερώτηση για την ανεργία των νέων. Και εκεί γίνεται μια συζήτηση. Τι θα γίνει με την εγγύηση για την νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν έχω κατασταλαγμένη άποψη, αλλά πριν να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και πώς να προχωρήσουμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι στο παρελθόν. Έπιασαν τόπο. Έχετε καταλήξει σε κάποια αξιολόγηση και για τη χώρα σας, ας πούμε πιάνουν τόπο τα κονδύλια εκεί για την εγγύηση για την νεολαία και πού χωράνε βελτιώσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιονκέριος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς για την παρουσία τους και για την παρουσίαση του προγράμματός τους. Φαντάζομαι ότι θα είναι ιδιαίτερο να αναλαμβάνεις προεδρία τόσο νωρίς μετά την ένταξή σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια για αυτό το βαρύ έργο που σας περιμένει, γιατί είναι βαρύ ε, λόγω όλων αυτών που ήδη ακούσαμε και αναφέρετε κι εσείς. Πρώτη ερώτηση. Έχετε καμιά ιδέα ποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σαφή εντολή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο διότι για μας αυτό έχει σημασία. Και φυσικά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα κονδύλια που είναι στη δική μας αρμοδιότητα. Από καιρού εις καιρών ε, αποκομίζουμε την εντύπωση ότι το Συμβούλιο αδιαφορεί λίγο για τη συναπόφαση. Ενώ για μας η συναπόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική για το κοινωνικό ταμείο. Κάτι άλλο που πάλι έχει σχέση με τα οικονομικά. Χάρηκα πολύ αυτό που είπατε για την ε, υλοποίηση του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Αλλά πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Χρειάζονται και χρήματα για να αρχίζει η εφαρμογή ε, ε, αυτής της εγγύησης και να έχει ουσία. Πώς θα πείσετε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να δείξουν κάποια προθυμία και να αφιερώνουν και κονδύλια, όχι μόνο στη δίκαιη μετάβαση και την πράσινη συμφωνία, αλλά και στα κοινωνικά προγράμματα. Και τελευταία ερώτηση, εγγύηση για τα παιδιά. Η Επίτροπος από την Κροατία κατά τη διάρκεια της ακρόασης της ε, αναφέρθηκε πολύ θετικά σε αυτό. Θέλουμε πραγματικά να στεφθεί με επιτυχία αυτή η εγγύηση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε γνωστή και σαφή χρηματοδότηση από την αρχή του PDP. Ξέρω ότι όλες οι ερωτήσεις που κάνω έχουν σχέση με χρήματα. Τι να κάνουμε, το χρήμα κινεί ε, το μάτιο του το ε, κόσμο. Ο κύριος Πισλάρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Υπουργοί, θέλω να σας συγχαρώ για το φιλόδοξο πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε. Χαίρομαι που αναφερθήκατε σε πάρα πολλά κομβικά ζητήματα για την κοινωνία μας και εξ ονόματος της ομάδας Renew Europe ε, στην Επιτροπή μας ε, θέλω να σε ευχηθώ καλή τύχη ε, για τις συζητήσεις που θα κινήσουν και καλή επιτυχία οι δυνατώσεις περισσότερες. Η κινητικότητα, η ισορροπημένη κινητικότητα είναι πολύ σημαντική για να υπάρχει συνοχή και ισορροπημένη ανάπτυξη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνετε ε, όμως όταν μεταφράζεται αυτό σε βαριές σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί υπάρχουν κάποιοι που περιμένουν 15 χρόνια ε, νομοθεσία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε νέα νομοθεσία για το συντονισμό ε, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, των αντίστοιχων ε, κανονισμών που έχουν οδηγηθεί σε εμπλοκή οι ψηφιακές λύσεις πραγματικά είναι η απάντηση ε, και είναι σημαντικό να προωθήσουμε την ψηφιακή εποχή για να ε, δίνουμε και να προτείνουμε καλύτερες λύσεις στους πολίτες. Στο κέντρο πολίτης πρέπει πάντα να βρίσκεται. Ε, τι πιστεύετε λοιπόν για αυτά τα στοιχεία και για τον κανονισμό 883 και την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Δεύτερον, ο δικό χάρτη προ μια κοινωνική Ευρώπη. Τον έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πρόγραμμά σα είπατε ότι θα δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για την εκρίζωση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού των πιο ευάλωτων, που είναι τα παιδιά, ε, ε, κάποιε ευάλωτε ε, ομάδε και περιθωριοποιημένοι Ρωμά. Με τη στέγη τι γίνεται. Κάναμε πρόσφατα μια συζήτηση για την κοινωνική στέγαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα της στέγης, θα το βάλετε ε, στο δικό σας πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή τύχη η κυρία Λάγκεντζίπεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί Υπουργοί, θα ήθελα καταρχά να σας πω ότι με χαρά άκουσα το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας σας. Ίσες ευκαιρίες, προστασία ε, ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ε, και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πολύ ελπιδοφόρα αυτά που διάβασα, ότι θα δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στην εκρίζωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των πιο ευάλωτων ομάδων. Παιδιά και άτομα με αναπηρίες. Και χαίρομαι που προγραμματίζεται και σχετική διάσκεψη για ε, τα άτομα με αναπηρίες και τη σύμβαση του ΕΟΑ και το, για τους περιθωριοποιημένους ΡΟΠΑ. Θέλω να σας ρωτήσω, τι κάνετε με τους αστέγους, αυτό σας απασχολεί, το θέμα το έχετε στο πρόγραμμά σας. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δρόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλεισμένοι ε, από κάθε δικαίωμα ανθρώπινο και αξιοπρέπεια. Στην πρώτη συζήτηση για τη στέγη στην ε, ε, Ολομέλεια ζήτησα από την Επίτροπο να προτείνει στρατηγική και τα κράτη-μέλη να κάνουν στρατηγική για τους αστέγους με μέτρα και προδραστικά αλλά και αντιμετώπισης για να ε, σταματήσει αυτή η απαράδεκτη στέρηση δικαιωμάτων των αστέγων. Ελπίζω στο Συμβούλιο να το προωθήσετε και εσείς αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζωμέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, σας ακούσαμε να μιλάτε για την ισότητα των φύλων, για τα δημογραφικά θέματα. Είναι πολύ σοβαρά. Μιλήσατε και για την ποιότητα της απασχόλησης και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις αποσπάσεις εργαζομένων ή να δούμε τι θα γίνει με τον συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων στην Ευρώπη. Ίσως να μας δώσετε κάποια στοιχεία, θα έλεγα, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις αδυναμίες του μηχανισμού λήψεως αποφάσεων στην Ευρώπη θα προωθήσετε ε, περισσότερο την κυριαρχία ε, των κρατών μελών στον τομέα αυτό ή κάτι άλλο. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργούνται επίσης και από την πολιτική λιτότητα και ξέρω ότι στη δική μου χώρα επηρεάζεται άμεσα το κοινωνικό σύστημα. Και ποια είναι η πολιτική σας για τη συμπερίληψη των εργαζομένων ε, μεταναστών που πολλές φορές γίνεται εις βάρος των γηγενών ε, και οδηγούμεθα έτσι σε συστήματα δουλείας ουσιαστικά. Και θα ήθελα να μάθω επίσης και τι γίνεται και με το λεγόμενο κοινωνικό dumping στα πλαίσια των αποσπασμένων εργαζομένων. Επιτέλους θα πρέπει η οικονομία να υπηρετεί τους πολίτες και όχι το αντίθετο. Πότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπηρετήσει τους λαούς που την αποτελούν. Κύριε Κύριε Υπουργέ κυρίες ε, και κύριοι. Παρουσιάσατε πολύ φιλόδοξα προγράμματα. Αναφέρατε και τις πραγματικότητες. Ο χρόνος όμως ε, εφαρμογής ε, δεν είναι πολύς. Έχει περάσει ένας μήνας ήδη και μετά θα έρθει και η Γερμανική Προεδρία. Οπότε δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος και η αρχή είναι δύσκολη γιατί έχουμε και την αρχή του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος. Έχω πάντα την εντύπωση πως ε, η Προεδρία αυτό είναι η Κροατική ή η Γερμανική. Δηλαδή εντάξει γίνονται οι συζητήσεις εις ε, βάθος αλλά πότε θα δράσουμε πιο συγκεκριμένα. Έχουμε πολλές προκλήσεις και δεν κάνουμε αρκετά και αντιλαμβάνομαι πως ε, κάθε κρατος μέλος που έχει την Προεδρία έχει κάποιες ε, φιλοδοξίες, ε, θέλει να επιτύχει κάποιους στόχους, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στα δημογραφικά προβλήματα που πρέπει να τα δούμε μακροπρόθεσμα. Πώς θα υπάρξει μια μακροπρόθεσμη εγγύηση. Υπάρχουν ε, πράγματα, τα είπαν και οι συντονιστές, ε, η εγγύηση για τους νέους, ε, ο ευρωπαϊκός βασικός μισθός, πώς θα προχωρήσουμε. Μιλήσατε για διαβούλευση. Τι διαβουλεύεστε, υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο. για τον συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα, θέλετε να επιταχύνετε. Γιατί κάπου έχουμε κολλήσει. Όταν επίσης μιλάμε για έλλειψη εργασίας ε, των γυναικών. Ε, κάπως πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερως η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και εντάξει, η παθητικότητα μπορεί να έχει διαφορετικές αιτίες σε κάθε χώρα. Τι άποψη έχετε επίσης για τις εξελίξεις ε, στα ζητήματα κοινωνικών παροχών. Κύριος Βίλεμσεν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, και εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Έχω μία ερώτηση για το πρόγραμμά σας, γιατί εκεί πέρα λέτε ότι ευθυγραμμίζεστε με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και θα ενθαρρύνεται μια συζήτηση για τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Εμείς, όπως το βλέπουμε ως αριστερά, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Χαμηλή μισθή, ε, επισφαλείς ε, δουλειές και τα μπλοκάκια επίσης. Οπότε η άποψή μου είναι ότι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε αξιοπρεπή δικαιώματα για τους εργαζόμενους είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα όμως να ακούσω τις δικές σας τις απόψεις πιο συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, προκλήσεις. Μετά από τον πρώτο γύρο ερωτήσεων θα ακούσουμε και τις πρώτες απαντήσεις. Ε, ποιος θα ξεκινήσει. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Σας, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. i dijela Epsko vijeća koji vodimo pokušati odgovoriti na dio pitanja naravno, a drugi... Εξ ονόματος του Υπουργείου και του Συμβουλίου θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις μας αφορούν τα υπόλοιπα θα τα δει συνάδελφος. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω απαντήσεις στα θέματα τα οποία είναι στις δικές μου αρμοδιότητες και μετά η συνάδελφος θα δώσει τις υπόλοιπες απαντήσεις. Σχετικά... 19. Πρέτσινικ Σαρλ Μισελ Σχετικά με το ΠΔΠ και εδώ έρχομαι και στις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο πρόεδρος Σαρλ Μισελ ε, οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε εμείς ε, ως Προεδρία ε, να πω είναι ότι μια πρακτική που ακολουθείται όταν δεν υπάρχει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο ή σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Το πολιετές δημοσιονομικό στην παρούσα φάση λοιπόν δεν έχει επιληθεί, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια συνενετική λύση και στον τομέα αυτό που οι δυσκολίες είναι αρκετά μεγάλες. Αν δούμε το πώς έχουν εξελιχθεί μέχρι τώρα τα πράγματα, ανατομέα, νομίζω ότι θα χρειαστεί αναμονή, θα χρειαστεί χρόνος για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σχετικά πάντα με το πολιετές δημοσιονομικό, υπήρξαν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. Συν. Οι συζητήσεις και εδώ συνεχίζονται, αλλά καταλαβαίνετε ότι εξαρτάται απόλυτα από τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν για το πολιετές δημοσιονομικό. Αν δεν έχουμε ε, κάτι το παγιωμένο από πλευράς ε, ε, πι τότε είναι δύσκολο να προβλέψουμε οτιδήποτε για το κοινωνικό ε, ταμείο ΣΥΝ. Το κοινωνικό ταμείο έχει λειτουργήσει σωστά, έχει βελτιώσει ε, τις συνθήκες στον τομέα της παιδείας, στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και είχε επίσης και θετικές επιπτώσεις στη σύγκληση των κρατών μελών σχετικά με τον ελάχιστο μισθό. Ε, ήδη στις 14 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρώτο σχέδιο εγγράφου γύρω από τις κοινωνικές διαπραγματεύσεις που θα προηγηθούν του καθορισμού ενός ε, κοινωνικού ελάχιστου ε, μισθού. Ε, ο μηχανισμός αυτός σε επίπεδο κοινωνικό έχει πολύ μεγάλη σημασία 22 ε, από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια κάποια νομοθετική ρύθμιση γύρω από ένα ελάχιστο κοινωνικό μισθό. Συνεπώς λοιπόν θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος του εξαμήνου μας να κάνουμε βήματα προόδου τουλάχιστον σε επίπεδο Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ ε, έχοντας τουλάχιστον ορίσει το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, γιατί και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Συνεπώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες να σας μεταφέρουμε, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια πραγματική συζήτηση για την μορφή την οποία θα μπορούσε να έχει ε, το σύστημα του ελαχίστου μισθού, τον οποίο θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω λοιπόν στοιχεία για τον πιθανό συμβιβασμό ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα, ε, για τα κοινωνικά δικαιώματα σε επίπεδο πολιτικό ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις, μάλλον αυτό είναι ο τομέας στον οποίο γίνονται οι συζητήσεις ε, οι σημαντικές σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτού που λέμε κοινωνική Ευρώπη. Αυτό το επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών το οποίο έχει υιοθετηθεί ήδη από το 2017 με μια κοινή ε, δήλωση το 2017 επαναλαμβάνω θα πρέπει λοιπόν αυτό το ε, καθορισμένο επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων να υπάρχει και να γίνεται αναφορά σε αυτό σε όλες τις κοινωνικές ρυθμίσεις τις οποίες υιοθετούμε έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Σχετικά τώρα με τον κανονισμό το 883 ή καλύτερα την αναθεώρηση του κανονισμού 883 ήδη από την Φιλανδική Προεδρία συνειδητοποιήσαμε τη σημασία που έχει ο κανονισμός αυτός για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε λοιπόν ενημερωμένοι για την κατάσταση της συζήτησης αυτής. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά ελπίζουμε ότι σε συνεργασία και μαζί σας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση έτσι ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Η προσπάθειά μας λοιπόν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι να προχωρήσουμε σε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε να γίνει δεκτή η πρόταση της Επιτροπής. Καθορίζονται στα πλαίσια αυτής της πρότασης ορισμένοι κανόνες σε επίπεδο κινητικότητας, μεταφοράς δικαιωμάτων κτλ. Είναι κάτι το οποίο επίσης θα διασφαλίσει μεγαλύτερη, ε, θα έλεγα, ισότητα ανάμεσα στους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Τώρα για τις κοινωνικές διαπραγματεύσεις ε, και τον κοινωνικό διάλογο. Είναι σαφές ότι ενδιαφερόμεθα για τον κοινωνικό διάλογο και υποστηρίζουμε τον κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ευρώπη. Είναι, θα γίνει μια συνάντηση στις 23 του μηνός σε τριμερές επίπεδο και θα αντιμετωπιστούν θέματα όπως ε, τα χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων ε, και ε, οι κανόνες με τους οποίους θα προχωρήσει ο τριμερής αυτός διάλογος. Πιστεύουμε ότι ε, οι κοινωνικές διαπραγματεύσεις θα δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι ο κοινωνικός διάλογος και όπου έχουμε την δυνατότητα να τον προωθήσουμε θα το κάνουμε. Νομίζω ότι δεν έχω να δώσω κάποιες άλλες απαντήσεις ε, και θα ήθελα να περάσετε το λόγο τώρα στην συνάδελφό μου, την κυρία Μπεντιακόβιτς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω κι εγώ Λοιπόν, όπως έκανε και ο συνάδελφος, θα ομαδοποιήσω και εγώ τις απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όταν ε, σκεφτόμαστε στρατηγικά για το μέλλον των κοινωνικών πολιτικών θεωρούμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε ε, αποτελεσματικά στις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές και για τον λόγο αυτόν οι πολιτικές μας χρειάζονται μια συνέχεια και κάποια πρόοδο. Λοιπόν, για να έχουμε ένα σύστημα χρειάζεται να εργαστούμε στρατηγικά και συστηματικά. Και θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι προσιλωμένοι σε αυτόν τον στόχο. στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε την συνέργεια μεταξύ ε, οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και οι κοινωνικές αρχές, ε, τα κοινωνικά δικαιώματα να είναι στο επίκεντρο της ε, προσοχής μας. Όταν μιλάμε λοιπόν για κοινωνική προστασία ένας άλλος ε, σημαντικός ε, παραγόντας είναι οι εθνικές ιδιαιτερότητες και οι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Γι' αυτό παρακολουθούμε στενά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε τους επόμενους έξι μήνες όλες τις ε, πρωτοβουλίες που είχε ήδη ξεκινήσει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν το μέλλον της ε, κοινωνικής Ευρώπης και την ενίσχυση της ε, κοινωνικής Ευρώπης. Θα εστιάσουμε επίσης σε μια πιο δικαίη μετάβαση στην ισότητα των φύλων και στην διαφάνεια των μισθών. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα. Εδώ θα εστιάσουμε στην ε, συνεπή εφαρμογή όλων των στοιχείων του κοινωνικού πυλώνα γιατί θεωρούμε ότι η εφαρμογή των αρχών που περιέχονται σε αυτά τα έγγραφα είναι πάρα πολύ σημαντική όταν μιλάμε για το μέλλον της ε, κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη σήμερα είναι μοναδική. Ευημερία, δικαιοσύνη και βιώσιμο μέλλον είναι στόχοι που είναι εξίσου σημαντικοί. Επίσης γνωρίζουμε ότι ο στόχος μας αλλάζει γρήγορα. Υπάρχουν λοιπόν ε, νέες προκλήσεις ε, αλλά και νέες δυνατότητες. Θα εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή μας σε όλες τις προτάσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλες μας οι προσπάθειες θα είναι προς την κατεύθυνση της περαιτέρω εξέλιξης μιας κοινωνικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις ε, ερωτήσεις σας αφορούσε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και σας ευχαριστώ γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό ειδικά δεδομένου του ότι παρά την θετική πρόοδο εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος φτώχειας ε, και κοινωνικού αποκλεισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για παιδιά, μειονότητες, ε, μετανάστες, ανάπηρους. Όλες αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση, στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες. στην αγορά εργασίας. και βεβαίως Το ίδιο ισχύει και για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν πιο προστατευμένοι στην προηγούμενη κρίση. Οι κοινωνικές επενδύσεις και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό θεωρούμε ότι ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι η πηξίδα, ο μπούσουλας που θα μας κατευθύνει προς τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Και αποτελεί και έναν πάρα πολύ σημαντικό στόχο για να επιτύχουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις αγοράς-εργασίας, όπως ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της στόχιας ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, και η ανισότητα. Ένα άλλο ερώτημα τέθη όσον αφορά τις εργατικές κατοικίες ε, και τους άστεγους. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό. κατάσταση με την στέγαση και εδώ περιλαμβάνονται και οι άστεγοι είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλά κράτη-μέλη Και πρέπει να λυθεί με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πρέπει να υπάρξει πρόληψη και στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα συλλογής και παρακολούθησης δεδομένων και να περιλάβουμε περισσότερους ενδιαφερόμενους στην ε, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει λοιπόν να βρούμε περισσότερους πόρους, να μιλήσουμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε βέλτιστες ε, πρακτικές καθώς αυτοί οι παράγοντες οπωσδήποτε ε, τελικά θα μας οδηγήσουν σε αλλαγές. Οπωσδήποτε θα το δούμε αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που ετέθη αφορά το θέμα των ατόμων με αναπηρίες. όπως είπα εμείς ε, εστιάζουμε στα ζητήματα αυτά την Ευρωπαϊκή ημέρα ατόμων με αναπηρία και την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία και πρέπει ακριβώς ε, να προστατεύσουμε αυτά τα άτομα και να έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα και δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή. Τονίζουμε λοιπόν την ανάγκη να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση για να τονίσουμε τα ζητήματα αυτά σε διάφορους τομείς της πολιτικής. Βεβαίως η δουλειά μας δεν σταματά εδώ θέλουμε να φροντίσουμε όλα τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και θα εργαστούμε για την εφαρμογή της ε, σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητά μας. Οι πληροφορίες που έχουμε από τα στατιστικά στοιχεία και τα δεδομένα από την δημόσια διαβούλευση είναι σημαντική συνεισφορά και βεβαίως θα μας ε, βοηθήσουν στις μελλοντικές μας δραστηριότητες. Εδώ πρέπει να μπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια συστηματική προσέγγιση. Οπωσδήποτε θα γίνει μια διάσκεψη για να αξιολογήσουμε τις αναπηρίες και να χρηματοδοτήσουμε τις ενός ατόμων με αναπηρία. Η δε διάσκεψη θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της ε, σχετικής σύμβασης του ΟΗΕ τα ζητήματα χρηματοδότησης των ενώσεων αυτών, την αξιολόγηση των αναπηριών, την θέση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και ελπίζουμε να ξεκινήσει μια εύρια συζήτηση για το θέμα αυτό και να ενθαρρύνουμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των κρατών μελών. Υπήρχε επίσης ένα θέμα για την εγγύηση για τα παιδιά. Εδώ πέρα απαιτείται η πολιτική βούληση. Οι κατευθυντήριες γραμμές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ισχυρή δράση για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, καλύτερη διασύνδεση των ταμείων. Αυτά είναι στοιχεία που είναι αναγκαία για να ενισχυθεί αυτό το σύστημα. Η έγκαιρη παρέμβαση επίσης έχει σημασία πέρα από το, ε, την εξοικονόμηση χρημάτων έχει μεγάλη σημασία για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που είναι ένας φαύλος κύκλος. Αναμένουμε λοιπόν την διάσκεψη αυτή που θα γίνει στο τέλος της πρώτης φάσης στις 17 Φεβρουαρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις θα μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την συζήτηση αυτή. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βελτιωθεί το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και πρέπει να συνεχίσουμε την καταπολέμηση της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών. Αλλά πρέπει να υπάρχει και προστασία, πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση και στέγαση για όλα τα παιδιά που κινδυνεύουν. Αν ε, το σημείωσα σωστά υπάρχει και ένα ερώτημα για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Όπως είπα στην αρχική μου ομιλία, η συμπεριληψή των γυναικών ε, στην αγορά εργασίας είναι βασικό ε, στοιχείο οικονομικής ανεξαρτησίας ανδρών και γυναικών και θα οδηγήσει σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό ο στόχος μας είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να καθοριστεί ο ρόλος των θεσμικών οργάνων, να παρακολουθούνται τα στατιστικά δεδομένα, να έχουμε στοχευμένες στρατηγικές για αυτό το ζήτημα και τέλος να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων που έχουν αναλυθεί για να λυθεί αυτή η πρόκληση. Μετά έχουμε ζητήματα που αφορούν τις δημογραφικές προκλήσεις. Τα είπα αυτά στην αρχή μου ομιλία, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω σχεδόν Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν ε, σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουν διάφορες ε, δημογραφικές προκλήσεις. Το να ξεπεράσουμε αυτές τις ε, προκλήσεις έχει μεγάλη σημασία για να ενισχύσουμε την κοινωνική σύγκληση και την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω πως η Κροατία ήταν αυτή η οποία προώθησε αυτό το θέμα. Αναγνωρίσαμε λοιπόν στη χώρα μας ότι είναι πρόβλημα και έχει μπει στο στρατηγικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το επόμενο πενταετές ε, πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτό το θέμα. και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε εις βάθος. Οπότε και τις αρνητικές ε, δημογραφικές τάσεις αλλά και πολιτικές που θα βελτιώσουν την ζωή των πολιτών μας. αλλά βεβαίως και η δυνατότητα να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματική ζωής θέλουμε να εστιάσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, στους ανθρώπινους πόρους ε, και στις μελλοντικές πολιτικές της Ένωσης, οι οποίες πρέπει να εστιάσουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών τάσεων. Και βεβαίως ε, για ίση οικονομική ανάπτυξη όλων των ε, κομματιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε πλήρη επίγνωση όλων αυτών των προβλημάτων και όλων αυτών των στοιχείων που μεταφράζονται επίσης και ε, με τις δημογραφικές εξελίξεις και οπωσδήποτε βαρύνουν την ε, οικονομία μας θα ανοίξουμε μια ευρύτατη συζήτηση για αυτό το θέμα. Για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, ε, εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών για να μπορέσουμε στη συνέχεια να εκρίνουμε συμπεράσματα. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η πρώτη απάντηση στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Έχουμε και δεύτερο γύρο τώρα ερωτήσεων. Σύντομα να διαβάσω τα ονόματά σας και η κυρία Μπίσοφ.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 Αρχίζει και πιέζει λίγο χρόνος. Α, και η κυρία Λίζη και ο κύριος Πάτεν. Ωραία. Έλεγα ότι έχει αρχίσει και πιέζει λίγο χρόνος. Θα πρέπει να βάλουμε κανόνες. 1,5 λεπτό για την ερώτησή σας, ο καθής. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Αρχίζουμε από την κυρία Τόμς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ για τις παρουσιάσεις σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που στις προτεραιότητές σας έχετε προβλέψει και την ισχυρή Ευρώπη. Για να είναι η Ευρώπη ισχυρή όμως και να υπάρξει, θα πρέπει να είναι και τα, κάθε κράτος μέλος ισχυρό. Ξέρουμε ότι η αλυσίδα είναι ισχυρή όσο είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που δεν είναι οι πιο ανταγωνιστικές. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διάφορα ταμεία, μεταξύ αυτών το Ταμείο Συνοχής. Ε, ακούσαμε και για το Κοινωνικό Ταμείο. Εσείς θα είστε αρμόδιοι για τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ελπίζω πάρα πολύ η θέση σας να είναι ότι δεν μπορούν να μειωθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ε, στο βωμό του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Ερωτώ λοιπόν Πρώτα απ' όλα για το δημογραφικό. Ε, χαίρομαι που έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτό το πρόβλημα οξύνεται όλο και περισσότερο. Οι λύσεις όμως ποιες είναι. Θα ήθελα να ακούσω κάποια σχετικά. Θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε απτές λύσεις και προτάσεις για το αυξανόμενο δημογραφικό πρόβλημα. Τι μπορούν να κάνουν εδώ οι ευρωπαϊκές πολιτικές για να το αντιμετωπίσουν. Το ξέρω ότι αυτό είναι κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και τελευταία ερώτηση, τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι οι νέοι από χώρες όπως είναι η Κροατία, η Σλοβενία, η πατρίδα μου, δεν θα αναγκάζονται να ξενιτεύονται, να πηγαίνουν σε δυτικές χώρες οι πιο ανεπτυγμένες ο κύριος Κάσα και να ετοιμάζεται ο επόμενος ομιλητής, ομιλητρία. Ευχαριστώ τους υπουργούς που ήρθαν για την παρουσία τους, για την παρουσίασή τους και τις λεπτομερέστατες απαντήσεις τους. Μαζί με τους άλλους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή είμαι αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και επιτρέψτε μου να επανέλθω, είναι πολύ σημαντικό, βοηθάει εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Είμαι πολύ σίγουρος ότι τα ξέρετε αυτά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επενέσω τη διαπραγματευτική ομάδα, την Κροατική, για την επικοδομητική στάση στις πρώτες τεχνικές συνεδριάσεις. Πρώτη συνεδρίαση έγινε αυτή την εβδομάδα. Το επικοδομητικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας που πριτάνευσε εκεί για τα ε, προβλήματα που πρέπει να λυθούν και με ταχύτητα. Έχω όμως ανησυχίες. Ανησυχώ Στη Φιλανδική Προεδρία είχαν έρθει κάποιες προτάσεις που κυκλοφορούσαν στο Συμβούλιο για περικοπές του Κοινωνικού Ταμείου. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ο Ντένις, ανησυχώ πολύ προσπαθούν να αποσπάσουν ακόμα περισσότερα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ προς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Και θυμίζω ότι αν υπάρξει γενναία περικοπή στο ε, ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα έχει τεράστιες συνέπειες στα κράτη-μέλη. Υπάρχει και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ε, υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ ε, Εντό των διαπραγματεύσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι το Κοινοβούλιο είναι στεναρά κατά αυτών των συμπεριλήψεων στι διαπραγματεύσει. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε τη βοήθειά σα για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα στι διαπραγματεύσει. Η κυρία Λοραντινέλη και να ετοιμάζεται η κυρία Ζελεύσκα. Ευχαριστώ η προτεραιότητά σας περιλαμβάνουν και την προσπάθεια διεύρυνσης προς τις αλβαλκανικές χώρες. Είναι απαραίτητο όμως να προστατεύσουμε κάποια επίπεδα ζωής και κάποια κοινωνικά δικαιώματα για να καλύψουμε και το τραυματικό παρελθόν των λαών αυτών των χωρών. Η αλήθεια είναι ότι η ένταξη μαζική των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 90 δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα ε, στην εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη τα οποία είχαμε κάνει τότε. Τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε τέτοιου είδους φαινόμενα να μην εξακολουθούν να ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. κυρία Ζαλεύσκα είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ ε, τους υπουργούς. Έχουμε και εμείς επιφυλάξεις και ανησυχίες. Ενδεχομένως πόροι από το Ταμείο Συνοχής να χαθούν και να πάνε σε αυτή την περίφημη πράσινη μετάβαση. Και τώρα θα πρέπει να σκεφτούμε πού θα βρούμε φρέσκο χρήμα. Ε, όχι να αρχίσουμε τις περικοπές στα διάφορα υπάρχοντα ταμεία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβληματιστεί. Ωραίο το πρασίνισμα, αλλά θα πρέπει να βρούμε και χρήματα για να το κάνουμε αυτό. Ε, να δούμε και ποια χρήματα θέλουμε να αφιερώσουμε σε ποιους σκοπούς μας. Αναφέρατε εσείς κάποιες προτεραιότητες, οπότε είναι σημαντικό κάπως να τα ιεραρχήσουμε αυτά τα πράγματα και να καταλάβουμε ποιο είναι σημαντικότερο και ποιο λιγότερο σημαντικό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να έχουμε σωστή χρηματοδότηση. Υπάρχουν κάποια μεγάλα έργα, ας πούμε, ε, για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού στη χώρα μας. Όλα τα σχολεία τώρα στη χώρα μας έχουν ευρυζωνικότητα. Έχουν γρήγορο διαδίκτυο, μετεκπαιδεύονται οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί και τώρα δουλεύουμε σε άλλα project για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους που κινδυνεύουν από τον ψηφιακό αποκλεισμό και απειλούνται. Και έχουν ξανακάτσει στα θρανία για να μάθουν. Έχουμε μια στρατηγική στη χώρα μας και μπορούμε να δείξουμε ε, τι εστί διαβίου μάθηση και πώς μπορούμε αυτή να την προωθούμε. Και φέρνει και αποτελέσματα. Αντίστοιχους οργανισμούς επίσης έχουμε. Η πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια και δίνει το λόγο στον επόμενο μιλήτη, ο κύριος Ντάνιελσον. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς για την παρουσίαση της ε, Προεδρίας. Εγώ είμαι μέλος της ομάδας σοσιαλιστών και δημοκρατών και επιμένω πάρα πολύ στην κοινωνική Ευρώπη, στις συνθήκες εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και χαίρομαι που η Κροατική Προεδρία ακριβώς αναφέρεται στη σημασία του ε, Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή την προτεραιότητα. Επίσης χαίρομαι που τονίσατε πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικέ συμβάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε μια δίκαιη, βιώσιμη Ευρώπη και για να γίνει αυτό πρέπει να βασιστούμε στους κοινωνικούς εταίρους. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ η πολιτική μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλο σημαντικός κλάδος πολιτικής είναι η περιβαλλοντική, γιατί επηρεάζει την ευημερία και την ευζοία των εργαζομένων, των πολιτών. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν έκανε λόγο για την κοινωνική Ευρώπη, είπε ότι Κάθε ευρώ που επενδύουμε ε, αυγατίζει και γίνονται δύο ευρώ. Ε, εκεί. Ε, ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα επενδύουμε, πώς εργάζεται ο κόσμος, να μην υπάρχουν προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά και υγιές. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια στρατηγική για το περιβάλλον εργασίας, όχι για το περιβάλλον, για το χώρο εργασίας, για το πώς δουλεύει ο κόσμος, για να έχουμε ένα συνολικό όραμα, μια συνολική θεώρηση, να αποφύγουμε τις επαγγελματικές νόσους και τις ψυχικές νόσους και τα ψυχολογικά προβλήματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χόμς και να ετοιμάζεται η κυρία Φεράντης, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους υπουργούς της κορατικής Προεδρίας για τις προτάσεις τους. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημογραφικές αλλαγές δημιουργούν προβλήματα σε επίπεδο εδαφικό, σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο οικονομικό και υπονομεύουν την ισότητα των ευκαιριών και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με ικανοποιητικό τρόπο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μηχανισμούς οι οποίοι να βοηθήσουν τις περιοχές οι οποίες θα υποφέρουν και από τη μετανάστευση των νέων, την αποχώρηση των νέων από ορισμένε περιοχές και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ικανοποιητικού επίπεδου θέσεις απασχόλησης. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα στη δική μου χώρα τα οποία έχουν λειτουργήσει θετικά και τα οποία θα μπορούσαν να εξαχθούν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την δημογραφική πρόκληση. Ε, θα ήθελα να μάθω λοιπόν τι μέτρα θα χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να αυξήσετε ε, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες τις οποίες θα έχουν οι νέοι στις περιοχές της υπαίθρου και να υπάρξει η διατήρηση του συστήματος, ε, θα έλεγα, βιωσιμότητας και του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ορισμένες από τις ερωτήσεις έχουν ήδη τεθεί, αλλά θα πρέπει να τις υπογραμμίσω. Ε, ήδη την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την πρότασή της τη γνωστή ως Green Deal για μια οικονομία η οποία θα είναι ε, οικολογικά ουδέτερη και γι' αυτό ε, νομίζουμε ότι αυτό το οποίο ελείπει στην πρόταση αυτή είναι η λεγόμενη κοινωνική διάσταση ε, της, ε, του πράσινου αυτού προγράμματος του Green Deal. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν εάν η Κροατική Προεδρία λαμβάνει υπόψη της ε, στις προτεραιότητες της και την κοινωνική διάσταση του Green Deal. Ήδη από την Φιλανδική ε, Προεδρία είχε τεθεί το θέμα της ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανοποίηση των διαφόρων τμήματων που συναποτελούν την κοινωνία είναι κάτι το ζωτικό για τη σωστή ανάπτυξη της Ευρώπης. Και υπάρχει επίσης και το ένα άλλο επιμέρους θέμα που είναι η ψυχολογική υγεία ε, στο χώρο εργασίας, στο εργασιακό περιβάλλον. Έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια κάποιες μορφές χειροτέρευσης της ψυχολογικής υγείας. Ε, υπάρχουν προβλήματα με παθολογίες οι οποίες χαρακτηρίζουν πάρα πολλούς εργαζομένους. Είναι κάτι το οποίο είναι στις προτεραιότητές σας και αν ναι με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσετε. Η κυρία Λενουάρ και μετά η κυρία Μάξοβα. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ τις κυρίες και κυρίους υπουργούς. Σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανέπτυξε τον προηγούμενη εβδομάδα τον οδικό χάρτη για την κοινωνική Ευρώπη. Κανένας δεν θα πρέπει ε, να αγνοηθεί στον τομέα της υγείας και σε σχέση μάλιστα με τον καρκίνο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι το βασικός παράγον θνησιμότητας και των 50% των ασθενειών από καρκίνο οφείλονται συνδέεται με κάποιο τρόπο με την εργασία. Έχουν υπάρξει επίσης αποδεδειγμένες αυξήσεις στο καρκίνο του στήθους της γυναίκες οι οποίες εργάζονται ε, σε νυχτερινές βάρδιες. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Θέλετε να πάρετε κάποια μέτρα, θέλετε αυτό το πρόγραμμα για την καταπολέμηση του καρκίνου να καταστεί σημαντικό και στον τομέα της εργασίας. Η κυρία Μάξοβα και μετά η κυρία Σεμέδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ευχαριστώ και τους υπουργούς που μας παρουσίασαν ε, την Κροατική Προεδρία. Όπως είπε και μια συνάδελφος, δεν βλέπω ούτε εγώ πολύ συγκεκριμένες ιδέες. Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική πολιτική και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή χρηματοδότηση. Το είπε μια συνάδελφο προηγουμένω. Μας λέτε ότι ο πληθυσμό γυράσκει και έχετε δίκιο. Είναι η Ευρώπη έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την ε, πρόκληση. Πρέπει να είναι βιώσιμα τα κοινωνικά συστήματα, όχι μόνο σε κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προτεραιότητα εδώ, κατά την άποψή μου, είναι να ε, δοθεί ε, συνέχεια στον κανονισμό 883 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα, θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσατε να αγωνιστείτε να διατηρηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, παρόλο ε, που υπάρχει κίνδυνος και απειλείται αυτό το ταμείο να γίνει και να απορροφηθεί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Επίσης χαίρομαι για όσα είπατε για τα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και έγκριση της αναπηρίας. Καλό είναι να μας δώσετε και συγκεκριμένα όμως συμπεράσματα για το πώς ε, να βοηθηθούν ε, η ανάπηρη, να υπάρχει μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπήρου ενιαία ή ενιαίο σήμα για τα διόδια πανευρωπαϊκά κτλ. Η κυρία Σεμέδο. Και ο κύριος Αλαβάνος Νικολάου παρακαλώ να ετοιμάζεται. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την Υπουργό Μπεντέκοβιτς και έχει να κάνει με την διαρροή εγκεφάλων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, το δημογραφικό, ε, στην Προεδρία σας και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την κυκλοφορία των εγκεφάλων, όχι διαρροή εγκεφάλων. Αυτό τι σημαίνει. Πώς θα ήταν λύση αυτό και θα απαντούσε στη διαρροή εγκεφάλων, η κινητικότητα των εγκεφάλων δηλαδή και πώς θα δουλέψουν το κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερη ερώτηση προς τον Υπουργό ε, Αλάντροβιτς. Αναρωτιέμαι Ποια είναι η θέση των ε, ανατολικοευρωπαϊκών κρατών για την ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Εσείς πώς προσπαθείτε να τους πείσετε να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή που να είναι και αξιοπρεπές αυτό το εισόδημα για να μπορεί κανείς να ζει. Ο κύριος Αλαβάνος Νικολάου και να ετοιμάζεται ο κύριος Σαλίμπα. Ευχαριστώ. Ε, σε ολόκληρη... Θα μιλήσω στα ελληνικά. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόστηκαν από όλα τα κράτη-μέλη συγκεκριμένε πολιτικέ κατευθύνσει, οι οποίε έχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επί παραδείγματι, ενισχύθηκε με κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλε τι χώρε η ελαστική απασχόληση. Φτάνει το 1 τρίτο περίπου του, συνολικού, του, του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα πάρθηκαν μέτρα τα οποία διέλυαν τι συλλογικέ συμβάσει εργασία, όπω επί παραδείγματι ε, μέτρα που πάρθηκαν στην Ελλάδα με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης που εφαρμόζει η τωρινή για τη διάλυση της, των συνδικαλιστικών διαδικασιών έτσι ώστε να μην μπορούν τα συνδικάτα ουσιαστικά οργανωμένα να παρέμβουν και να έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τρίτον, προωθείται οι αλλαγέ, βαθιές αλλαγές στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικά το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης από κοινωνικό ζήτημα μετατρέπεται σε ιδιωτικό ατομικό. Θα πρέπει να το πληρώνει δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος από την τσέπη του περαιτέρω. Απέναντι σε αυτά τα τρία ζητήματα έχουν προκύψει πάρα πολύ μεγάλοι αγώνε σε μια σειρά από κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Ποια είναι η άποψη τη Κροατική Προεδρία για αυτά τα ζητήματα. Και ένα σχόλιο. Ε, μεγάλη αντιφατικότητα έχουν αυτά τα οποία μα παρουσιάσατε. Μιλάτε ότι υπάρχει έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Οι εκατοντάδε χιλιάδε νέοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι ε, απόφοιτοι πανεπιστημίων με μεταπτυχιακά προγράμματα, τι είναι. Δεν είναι ένα τέτοιο ε, δυναμικό το οποίο πηγαίνει από χώρα σε χώρα ψάχνοντα να βρει μια λύση και έρχεται αντιμέτωπο με τι ίδιε δύσκολε συνθήκε. Ή, και κλείνω με αυτό, το πώ θα λυθούν τα προβλήματα των παιδιών που είναι κοντά στη φτώχεια, όπω λέτε κι εσεί, όταν σε οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ένας άνθρωπο ο οποίο αμείβεται. Δεν μπορεί να ζήσει. Ο <clears throat> κύριο θέλω να ευχαριστήσω του υπουργού για τι τόσο λεπτομερεί εξηγήσει ε, που μα έδωσαν στι παρουσιάσει του και του εύχομαι καλή επιτυχία το επόμενο εξάμεινο. Μία από τι βασικέ προτεραιότητε τη Προεδρία σα είναι η ψηφιοποίηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στο να κάνει τα επόμενα βήματα και να γίνει πιο ανταγωνιστική για να δημιουργηθούν περισσότερε ευκαιρίε. Πέρα όμως από την ευελιξία και την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, η ψηφιοποίηση έχει φέρει και νέα προβλήματα και νέες δυσκολίες. Μεταξύ αυτών είναι κάτι που έχουμε δει και εμείς. Αυξάνονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας ε, πρέπει να εξορροπείται καλύτερα ο επαγγελματικό βίο με τον οικογενειακό και τον ιδιωτικό. Είναι νέε πραγματικότητε, νέα τα προβλήματα. Έχω λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αρχίσει ήδη να συζητεί τη σημασία ε, του να μπορείς να αποσυνδέεσαι, ε, να μην είσαι συνδεδεμένος 24 ώρες το 24ωρο σε ψηφιακό επίπεδο. Αυτό θέλουν οι εργαζόμενοι να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους. Ποιες είναι οι προθέσεις σας για αυτά τα σημεία. Και μια άλλη νέα πραγματικότητα που έχει εμφανιστεί είναι οι εργαζόμενοι στις ε, διαδικτυακές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δυστυχώς δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία εκεί και ρύθμιση και πολλοί θεωρούνται ε, αυτοπασχολούμενοι ε, με μπλοκάκια δηλαδή. Ποια είναι τα σχέδιά σας για τους εργαζομένους αυτούς. Η κυρία Μπίσοφ ε, να ετοιμάζεται, αλλά προηγουμένως ο κύριος ε, Μπεργκλέτς. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Σας καλωσορίζω και εγώ. Έχω μερικές ερωτήσεις. Θέλω να ακούσω τι προτίθεται να κάνει η Κροατική Προεδρία για να εντάξει την κοινωνική διάσταση ε, στην πολιτική της. Εκτός από την Πράσινη Συμφωνία, η κοινωνική διάσταση θα μπει και αλλού, ας πούμε, σε πολιτικές που έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας. Επίσης, σχετικά με την ε, δημογραφική αλλαγή, θέλω περισσότερο να ακούσω σε ειδικού τομεί ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών υπάρχει δυνατότητα να επηρεάσουμε τα πράγματα και τις αλλαγές. Γίνεται μια ευρύτατη συζήτηση, ξέρω ότι δεν είναι απλές οι λύσεις και τώρα ξεκινούν μόνο κάποιες διαδικασίες, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά όλων αυτών δεδομένων, πού θεωρείτε ότι χρειάζεται περισσότερο αλλαγή. Και μια άλλη ερώτηση, πολύ βασική ε, για την Επιτροπή μας. Πώς προτίθεστε να συνδυάσετε την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας χωρίς να αντικαταστήσετε και γυναίκες πολιτικές από κοινωνικέ πολιτικές. Η κυρία ε, Μπίσοφ και να ετοιμάσετε κυρία Λίζη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του προγράμματός σας με τόσες λεπτομέρειες και τόσο εκτενώς. Ακούσατε ότι εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης μας ενδιαφέρει ο κανονισμός για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Πάρα πολύ. Και εγώ η συγγήτρια θα ήθελα να το υπογραμμίσω ξανά. Διαπιστώσαμε, το ανέφερε ο κύριος υπουργό, ότι επί Φινλανδικής Προεδρίας είχε τονιστεί ε, η σημασία αυτού του κανονισμού για τους πολίτες. Το είχε καταλάβει η Φιλανδική Προεδρία. Φυσικά όλοι θέλουν να προσελκύουν εργαζόμενους με ε, προσόντα και δεξιότητες, αλλά όταν πρόκειται για επιδόματα και παροχές ε, κοινωνικές είναι πιο επιφυλακτικοί αλλά αυτός ο κανονισμός είναι στην καρδιά της κοινωνικής Ευρώπης και θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει αποτελέσματα ότι θέλει να ε, προωθήσει τη σωστή, τη δίκαιη κινητικότητα και να υποστηρίζει τους πολίτες της. Επειδή είμαι και από τους τελευταίους ομιλητές, θέλω να σας ρωτήσω σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 6 Ποια είναι η φιλοδοξία σας, θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα αριθμό. Έχετε πολύ ψηλέ φιλοδοξίες ότι θα κλείσει αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή χαμηλέ. Η κυρία Λίζη και να ετοιμάζει το κύριο Σπάτεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω λοιπόν τους δύο υπουργού Εγώ προέρχομαι από το Φριούλι Βενέτσια Τζούλια. Είμαστε γείτονες θα έλεγα. έχει ε, ένα μεγάλο χωριό στην περιοχή μου, λέγεται Μπούγε και εσείς έχετε μια ολόκληρη πόλη με το ίδιο όνομα στη δική σας χώρα, μοιραζόμαστε πολλά. Εσείς αναφερθήκατε σε ορισμένες προτεραιότητες ε, με επιφυλακτικό θα έλεγα τρόπο, αλλά με αρκετά συγκεκριμένο. Ε, θα ήθελα να δούμε εδώ ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι πολιτικές τις οποίες έχετε γενικότερα και θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο αυτά που θα σημειώσω τώρα. Τα προβλήματα των διαμεθοριακών εργαζομένων. Ε, τι προτάσεις επίσης θα κάνετε στον τομέα τον δημογραφικό. Ε, της οικογένειας ή θα δώσετε κίνητρα για μεγαλύτερη μετανάστευση. Ε, ίσως θα μπορέσαμε να δούμε τι θα κάνουμε και με τα Βαλκάνια για να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις. Σχετικά τώρα με την αηφόρο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους και κάθε πολίτη. Πώς ε, θα ε, προωθήσετε το ρόλο ε, των ουδέτερων διαμεσολαβητών, ενδιαμέσων. Ο κύριος Πάτεν, ο τελευταίος ομιλητής, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν την Κροατία σας εύχομαι ότι καλύτερο, είναι μια εξαιρετική χώρα, ε, είναι πανέμορφη, έχω πάει πολλές φορές και ένα από τα αγαπημένα μου μουσεία στον κόσμο, ε, το Μουσείο των Διαρριγμένων Σχέσεων ε, στο Ζάγκρεμπι είναι πολύ σημαντικό. Ίσως να κάνετε και ένα μικρό χώρο στο μουσείο σας για το Brexit. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα στα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε, τα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε στα πλαίσια αυτής εδώ της Επιτροπής. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση που θα δώσω το Ηνωμένο Βασίλειο από την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μια μακρά και υπερήφανη παράδοση ε, σε επίπεδο κοινωνικού μισθού, κοινωνικής προστασίας κτλ. Ε, θα προσπαθήσετε να λάβετε υπόψη σας και το παρελθόν του Ηνωμένου Βασιλείου ή θα ασχοληθείτε μόνο με τις δικές σας εμπειρίες. Λοιπόν, ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει. Ο κύριος Λάντροβιτς. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Κυρίως γιατί πιέζει και το πρόγραμμα έχουμε υποχρεώσεις και εγώ και η κυρία Υπουργός. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σύντομα. Λοιπόν, στον πρώτο γύρο δεν απάντησα στην ερώτηση για τον κανονισμό 883, την ε, δυνατότητε ψηφιοποίησης. Ε, σε γενικές γραμμές βεβαίως ε, στηρίζουμε την ανταλλαγή δεδομένων αλλά γνωρίζουμε το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν σε όλα τα κράτη-μέλη να περιληφθεί στην ανταλλαγή των δεδομένων. Τώρα μιλάμε για το ΕΚΤ ΣΥΝ και το Ταμείο Δίκαιης ε, Μετάβασης. Και ε, βεβαίω δεν θέλουμε να βλάψουμε το Ταμείο αυτό λόγω των άλλων ε, δραστηριοτήτων. Ο στόχος μας είναι στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις να έχουμε το έκτος ε, σημαντικό παράγοντα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σχέση με το πίδελταπή. και ε, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές ε, διαπραγματεύσεις θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον προγραμματισμό και για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ που θέλουμε να διατηρήσει την κοινωνική διάσταση μια διάσταση η οποία τρόπον την ανεβάζει το επίπεδο εκπαίδευσης, ε, κοινωνικής ένταξης ε, σε κάποια κρατημέλη. Στη διεύρυνση. Όταν ε, μιλάμε για διεύρυνση πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θεωρείται κάτι το θετικό και προσπαθούμε να περιλάβουμε τις χώρες οι οποίες δεν είναι ακόμα κράτη-μέλη στις δραστηριότητες ε, του Συμβουλίου ε, του άτυπου Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων που θα γίνει στο Ζάγκρεπ και στο περιθώριο εκεί θα έχουμε συναντήσεις με τους Υπουργούς Εργασίας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά στις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όταν μιλάμε τώρα για την ψηφιακή ένταξη και την ένταξη των ηλικιωμένων στην ψηφιακή κοινωνία, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Και βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο μας είναι ιδιαίτερο αγαπητό και θα προσπαθήσουμε να ε, το προωθήσουμε. Τώρα για την κοινωνική διάσταση του πράσινου deal. Θεωρούμε ότι και το Ταμείο Δικαιής Μετάβασης και το ΕΚΤΣΥΝ θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια κοινωνική διάσταση που θα έχει σχέση με το πράσινο deal και τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Γιατί με τον τρόπο αυτόν υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ε, ή από την άλλη κάποιες ανισορροπίες ε, στην αγορά εργασίας και μέσω κάποιων ταμείων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική διάσταση του Πράσινου Deal και να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές ε, του διαστάσεις. Η ψυχική υγεία τώρα στην αγορά εργασίας είναι η δεύτερη προτεραιότητά μας. Και όπως άλλωστε και η ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και θεωρούμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πιο ανοιχτά τα ζητήματα ψυχικής υγείας, ε, και το πώς ε, έχει η κατάσταση στην εργασία. Υπάρχουν πολύ γρήγορες αλλαγές στην αγορά εργασίας και αυτό επηρεάζει τις παραμέτρους ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Και θεωρούμε ότι μέσω της δεύτερης αυτής προτεραιότητάς μας θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε μια συζήτηση επί των ζητημάτων αυτών με σκοπό βεβαίως να ε, αποτελέσει η ψυχική υγεία μία από τις προτεραιότητές μας. Ένα άλλο θέμα αφορούσε ακριβώς την βιωσιμότητα των κοινωνικών συστημάτων στην Ευρώπη. Πρέπει να το συζητήσουμε τώρα και στο μέλλον Λοιπόν, όταν μιλάμε για την βυσιότητα αυτών των συστημάτων, οι καιροί είναι δύσκολοι. Από τη σκοπιά της ε, Προεδρίας μας πρέπει να εστιάσουμε ακριβώς στις ε, νέες αυτές ε, δεξιότητες για να υπάρξει προστιθέμενη αξία και να μπορέσουμε μέσω μακροπρόθεσμα να έχουμε μια οικονομία ευημερίας. Οπωσδήποτε Αυτό είναι και ζήτημα βιωσιμότητας. Ε, όσον αφορά τον βασικό μισθό, νομίζω ότι είμαστε ακόμα στη φάση που αναμένουμε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή μεταξύ της Κομισιόν και των κοινωνικών εταίρων. Και όπως είπα, ενθαρρύνουμε τον τριμερή κοινωνικό διάλογο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας για να γίνει ο κοινωνικός διάλογος κάτι το οποίο θα είναι μια κοινή προσέγγιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κάτι το οποίο θα έχουμε κατά νου βεβαίως, ε, για να μπορέσουμε να τον προωθήσουμε καλύτερα. Οπότε, όσον αφορά την αγορά εργασίας, νομίζω ότι απαντήσαμε σε όλες τις ε, ερωτήσεις πλην μίας ε, γιατί μου είπατε να βαθμολογήσω από το 1 έως το 6. Ε, υποθέτω το 6 είναι ο καλύτερος βαθμός, οπότε ε, ελπίζω οι προθέσεις μας να βαθμολογηθούν με 6. Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις σας. Οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν τις ε, δημογραφικές ε, προκλήσεις και αυτό με χαροποιεί. Γιατί ήδη στην αρχή μου ομιλία είπα ότι αναγνωρίζουμε ότι η δημογραφία είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο στην Κροατία, γενικώ σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Γι' αυτό χαίρομαι ε, που έχουμε την ίδια άποψη. Και για το ότι και εσείς ε, συμφωνείτε μαζί μας. καλό είναι το ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε κάποια θετικά βήματα. Όταν μιλάμε για δημογραφικά ζητήματα γενικώς. πρέπει να δούμε ότι δεν αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες τις ίδιες ε, προκλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε σύσταση κάνουμε πρέπει να είναι ευέλικτη. για να λάβει υπόψη τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες αλλά και την κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, αναφέρθηκε το θέμα της κινητικότητας των νέων σχετικά ειδικά η κινητικότητα νέων ε, δραστήριων νέων αυτό το ανέφερε και ο συνάδελφος εδώ οπότε εάν ε, θέλουμε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα αυτό πρέπει να έχουμε κατά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην έννοια της κινητικότητας, της ελεύθερης μετακίνησης και επίσης να λάβουμε υπόψη το ότι η κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών είναι και θεμελιώδες δικαίωμα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αφαιρέσει όλα τα εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων. Οπότε θα προωθήσουμε την κινητικότητα και τη μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η κινητικότητα ε, των ανθρώπων είναι μία από τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οπωσδήποτε θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στο να επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής θα εστιάσουμε στη δημογραφική σύγκληση. Θέλουμε να επιτύχουμε ένα ίδιο επίπεδο δημογραφικής ανάπτυξης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά κρατημέλη και πολλοί βουλευτές επίσης τόνισαν το ότι το θέμα αυτό τη δημογραφίας είναι ένα ζήτημα το οποίο μόλις αρχίσαμε να συζητάμε. Είναι λοιπόν αρμοδιότητα τη κυρία Σούιτσα, της Αντιπρόεδρου της Κομισιόν και η Κροατική Προεδρία σκοπεύει να ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση για τις δημογραφικές ε, προκλήσεις. Θέλουμε να προωθήσουμε πολιτικές οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, την ισορροπία της οικογενειακής ζωής ε, με την με τον εργασιακό βίο. Και δεδομένου το ότι είμαστε στην αρχή αυτή της διαδικασία. πρέπει να λύσουμε την κατάσταση. Είναι πάρα πολλέ οι προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συζήτηση η οποία θα γίνει θα πρέπει να είναι μια ευρυτάτη συζήτηση για να δούμε αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάποια συμπεράσματα. τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις για τους νέους στις περιοχές της Υπέθρου. Όπως επίσης ε, και πολλές ερωτήσεις ε, είχαν ε, σχέση με την έξοδο των νέων από κάποιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προτεραιότητα την οποία δίνουμε στους νέους στις περιφέρειες της Ευρώπης και στις περιοχές της Υπέθρου νομίζω ότι θα αναγνωριστεί από όλους σαν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπογραμμίσω ότι οι νέοι έχουν αρκετές δυνατότητες σήμερα τις οποίες δεν είχαν οι νέοι σε παλαιότερες περιόδους Υπάρχουν ε, πολλές ε, πηγές ενημέρωσης, ε, πολλές δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να πάρουν μέρος οι νέοι και στα πλαίσια των οποίων μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους ανεμπό. Οι νέοι σήμερα είναι αλήθεια ότι είναι πολύ πιο κινητικοί από ό,τι ήταν στο παρελθόν και σε επίπεδο σπουδών και σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης και σε επίπεδο ατυπικής ε, εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να προσανατολίσουν ε, τις επιλογές τους ε, και στις δυνατότητες οι οποίες παρέχονται. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι νέοι, ακόμα και σε μια σύγχρονη σημερινή Ευρώπη, είναι πάρα πολλές. Και οι δυσκολίες αυτές έχουν κυρίως σχέση με την απασχόληση. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά στοιχεία αβεβαιότητας ε, στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των νέων και αυτό είναι πιο οξυμένο στις περιφέρειες της Ευρώπης και στις περιοχές της Υπέθρο. Πρέπει να αυξήσουμε λοιπόν τις πιθανότητες εργασίας στις περιφέρειες αυτές τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ελπίζω να περιλαμβάνουν στοιχεία ε, προς την κατεύθυνση αυτή και θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να αποκριθούμε με πιο ικανοποιητικό τρόπο στις προσδοκίες των νέων. Μια δεύτερη προτεραιότητα είναι η ευαισθητοποίηση για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι με περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση και στα πλαίσια του Συμβουλίου Νεότητας ε, και Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και άλλα θέματα που συνδέονται ε, με την κατάσταση των νέων στις περιφέρειες, όπως επίσης και με τη λεγόμενη φυγή των εγκεφάλων, ένα παράγων ο οποίος μπορεί να παίξει θετικό ρόλο είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή των νέων φυσικά. Νομίζω ότι είναι ένα κλειδί για την ε, ε, καταπολέμηση του αποκλεισμού των νέων από την αγορά εργασίας. Και να προσθέσω επίσης εδώ κάτι που ξέχασα προηγουμένως και κλείνοντας την παρέμβασή μου, ε, ότι θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν σε ε, ένα από τα χαρακτηριστικά, τα πολιτιστικά της πρωτεύουσας της χώρας μου, του Ζάγκρεμ, το Museum of Broken Relationships, δηλαδή το Μουσείο των Διαρριγμένων Σχέσεων. εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατανοούμε την απόφαση αυτή και τη σεβόμεθα, αλλά είστε όλοι καλοδεχούμενοι στην χώρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας αξιότιμη προσκεκλημένη για την παρουσίαση ε, των προτεραιοτήτων της Κρατικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις των συναδέλφων που έδειξαν ακριβώς έτσι, ένα γνήσιο ενδιαφέρον το, το, και ειλικρινέ για τα θέματα που μας απασχολούν όλους. Καλή σας τύχη, είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμά σας και φυσικά θα συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να επανέλθω στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που ήταν η έγκριση της ημερήσιας διάταξης we all what Mr. Ε, ακούσαμε όλα αυτά που είπε ο κύριος Πάτεν για το Brexit. Το σκεφτόμουν. Θέλω να πω σύντομα κάτι διαδικαστικά. Πώς φτάσαμε ως εδώ. Στην επιστολή, αντί να έχουμε μια κανονική γνωμοδότηση. Επελέγει αυτή η μορφή γνωμοδότησης βάσει του άρθρου 56 του κανονισμού. Και όπως όλοι γνωρίζετε, αυτό που θελήσαμε στην αρχή ήταν να έχουμε κανονική γνωμοδότηση με σκιώδεις, συντάκτες, ε, τροπολογίες, όλη η διαδικασία, αλλά ε, ε, πίεζε τόσο πολύ το χρονοδιάγραμμα λόγω των εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Συμφώνησαν λοιπόν οι συντονιστές στις 24 Οκτωβρίου να επιλεγεί μια πιο ευέλικτη μορφή εργασίας που ήταν η επιστολή την οποία συνέταξαν οι ε, συντονιστές και ενέκρινε η Επιτροπή μας. Χάρη σε αυτή λοιπόν την επιλογή των ε, συντονιστών ε, καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στο σχέδιο γνωμοδότησης και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις λόγω αυτής της ευελιξίας η διαδικασία και δημοκρατική ήταν και απολύτως διαφανής. Παρόλα αυτά, αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση πριν την ψηφοφορία. Ουσιαστικά τώρα έχουμε δύο ε, δυνατότητες. Πρώτον, να κάνουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων σήμερα στις 11 ή λίγο μετά, εν πάση περιπτώσει στις 11 θα πάρουν το λόγο οι συντονιστές ή ένας από κάθε πολιτική ομάδα και ο κύριος Πάτεν που έθεσε το ζήτημα. Η δεύτερη δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε σήμερα μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων στις 2.30 ώρα το μεσημέρι με τους ίδιους ομιλητές, συντονιστές ή ένας που θα ορίσει κάθε πολιτική ομάδα και ο κύριος Πάτεν. Και μετά είτε να ψηφίσουμε μετά τη συζήτηση πρωί απόγευμα. So these are the two options. Αυτές είναι οι δύο δυνατότητες, στα δύο δεχόν. Εγώ θα προτιμούσα το πρώτο, το α. Anybody who would like to add something. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα να πείτε, ο κύριος Πάτεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε έχω κάποια σχόλια. Πρώτον, χαίρομαι και εκτιμώ ε, ε, την ευελιξία σας, που είναι και δύσκολο. Προσωπικά θα προτιμούσα το δεύτερο να συζητηθεί το μεσημέρι για να μπορέσουν να ενημερωθούν όσοι δεν γνωρίζουν το θέμα και δεν έχουν παρακολουθήσει. Τώρα είναι 11 και 5 έτσι κι αλλιώς. ε, μα, ε, ωραία, να αποφασίσουμε γρήγορα. Ε, προτιμώ το δύο, κύριε Άγιον Κέριος. Εγώ θα προτιμούσα το πρώτο. Αλλιώς θα σπάσει η ψηφοφορία, η ώρα της ψηφοφορίας και δεν ξέρω πόσοι θα είναι διαθέσιμοι για να ψηφίσουν το απόγευμα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν είναι επιλογές ένα και δύο, μόνο η πρώτη είναι. Ο κύριος Ράτκε, ευχαριστώ. Να ψηφίσουμε τώρα. Όλοι έχουμε πολύ σφιχτά προγράμματα. Και είναι πολύ σημαντικές οι ψηφοφορίε που μπαίνουν εμβόλυμα. Και δεν μπορούμε τώρα να περιμένουμε του συναδελφούς να τα ανατρέπουμε. Άλλος. Καλώ. Άρα επικρατεί η πρώτη ε, επιλογή. Αρχίζει τώρα η συζήτηση με τη σειρά των πολιτικών ομάδων. Θα μας πείτε ε, ποιος θα πάρει το λόγο, ο συντονιστής ή κάποιος άλλος που θα ορίσει η ομάδα σας. Ο κύριος Ράτκε πρώτος. We are launching the discussion, right? Κύριε Ράτκε, έχετε το λόγο για να μιλήσετε πριν τις ψηφοφορίες. Ο συντονιστής του ΕΛΚ. Ο κύριος Κάζα, μα γιατί να κάνουμε συζήτηση, να ψηφίσουμε θέλουμε εμείς. Μα αυτή ήταν η πρώτη επιλογή που είπατε ότι θέλετε. Μικρή, σύντομη συζήτηση πριν τις ψηφοφορίες για αυτό το θέμα που έθεσε το πρωί ο κύριος Ράτκε για το διαδικαστικό. Mr. Pislaro, please. Κύριος Πισλάρο. Εγώ κατάλαβα ότι αυτή είναι η επιλογή πρώτη. Όλοι αυτό καταλάβαμε. Εσείς κύριε Ράτκε τι καταλάβατε. Εγώ να ψηφίσω θέλω. Ναι, δεν ήταν αυτό το option A λοιπόν. Ήταν η συζήτηση και μετά ψηφοφορία. Να δηλώσω. Ωραία. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να, να γίνει το Brexit και εγώ θέλω να γίνει ψηφοφορία. Get the vote done. Αυτό είναι μια τρίτη επιλογή που προτείνεται, να μην γίνει καθόλου συζήτηση και να πάμε μέσα στη ψηφοφορία. Ωραία. Ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα τρία τώρα που προσθέσαμε ενδεχόμενα. Η κυρία Γιονγκέριος. Εγώ δίνω το χρόνο γόρευσής μου στο συνάδελφό που συνέταξε την επιστολή, τον κύριο Πιτζάρο. Mr. Okay, we'll start immediately, but ε. clear on that. Λοιπόν, θα αρχίσουμε αμέσω. Το καταλάβαμε όλοι. Θα κάνουμε μια πολύ σύντομη συζήτηση και μετά θα ψηφίσουμε. Ε, ο κύριος Πιζάρο, εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς συμφωνούμε απολύτως με την επιστολή και τη διατύπωσή της και ε, το περιεχόμενό της. Νομίζω ότι αντανακλά αρκετά πιστά τις συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή μας. Ανησυχούμε. Υπήρχε μια παλιά συμφωνία, τώρα έγινε μια νέα συμφωνία του Whitehall όπως ονομάζεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προστατεύσουμε τα ε, κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην εργασία όλα αυτά έχουν φύγει από το παράρτημα 4 και έχουν μπει στην πολιτική ε, δήλωση. Εκεί δεν έχουν την ίδια νομική ισχύ ε, ε, με την προηγούμενη κατάσταση όταν ήταν στο παράρτημα 4. Εάν δεν παραταθεί η μεταβατική περίοδος υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος και αυτό είναι στα τέλη του 2020 να έρθουμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση κατάσταση που θα ισοδυναμούσε ένα ε, άτακτο Brexit, χωρίς καμία συμφωνία, πράγμα που θέλαμε όλοι να αποφύγουμε. Η θέση μας λοιπόν ταυτίζεται με τη χτεσινή θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ανησυχούμε μόνο εμείς εδώ, ανησυχούν και άλλοι. Η βολή των Λόρδων. Αγωνιά. Το είδαμε χτες. Θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβουν έτσι ώστε να ε, λυθεί το πρόβλημα. Οποιαδήποτε μελλοντική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να παραγνωρίζει και να αγνοεί τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο κύριος Ράτκε. Δεν μιλήσατε. Από την ομάδα σας ποιος θα μιλήσει. Κοιτάξτε. Τι να πω τώρα, εγώ δεν ε, θέλω να φάω πολύ χρόνο γόρυψης. Συντάξαμε μαζί αυτή την επιστολή ως γνωμοδότηση και αυτή είναι η άποψή μας. Θα την υπερψηφίσουμε σήμερα. Δεν υπήρχε καμιά διαφωνία στο παρελθόν. Είναι γνωστά τα συμφέροντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής μας ναι, εγκρίνουμε την ε, πρόταση και θα χαρώ να γίνει και σύντομα αυτό, όσο γίνεται. Ο κύριος Πισλάρου, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μόνικα Σεμέντο για να μιλήσει εξ ονόματος της ομάδας Ρινιού. Ως σκιώδης εισηγήτρια της ε, ομάδας μου, ασχολήθηκα με την νεολαία. Υπάρχει ακόμα κάποια βεβαιότητα για τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι το Erasmus ε, Plus, Erasmus μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σημαντικό να παραμείνει η δυνατότητα ε, παράταση τη μεταβατικής περίοδου μετά το τέλος του 2020 για να αποφύγουμε τις καταστροφικές συνέπειες ενός άτακτου Brexit και για τους ανθρώπους και για τις εταιρείε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους, η κυρία Λάγκεν Ζήπεν, η κυρία Χάνσεν. Η κυρία Φίλιπς. Με το Brexit μπορεί να περισταλούν σημαντικά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από τη Συμφωνία Αποχώρηση έχει φαρηθεί η αναφορά σε ίσους κανόνες παιχνιδιού δεν είναι δεσμευτικά τα πρότυπα που προτείνονται. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος ε, να κάνουν περικοπές στα δικαιώματα των εργαζομένων οι Βρετανικές εταιρείες σε μια κούρσα προς τα κάτω με τις ευρωπαϊκές. Επίσης ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι δεν υπάρχει παράταση της μεταβατικής περίοδου. Είναι πάρα πολύ πιθανό ε, να μην προλάβει η κυβέρνηση να περάσει βρετανικούς νόμους για να αντικατασταθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, να ε, υπάρξει άτακτο Brexit χωρίς προστασία των εργαζομένων. Δεν μπορούν να πέσουν θύματα στο βωμό των ε, ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των εταιριών τους. Αυτή η συμφωνία αφήνει τη Βρετανία να κάνει ασίδωτη ό,τι θέλει. Θα πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τώρα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζαμέη, δεν ξέρω ποιος από την ομάδα σας, παρακαλώ. προσωπικά δεν συμφωνώ απολύτως με το ψήφισμα αυτό. Πολλές από τις επικρίσεις είναι ε, αδικαιολόγητες, ειδικά προς την κυβέρνηση. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση των Βρετανών. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι οι ανησυχίες σας είναι βάσιμες, είτε για τα κοινωνικά είτε για τα φορολογικά ζητήματα. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε τώρα, να παρεμποδίσουμε το Βρετανικό λαό να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει αποφασίσει. Και δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι όλοι από κοινού και ο Βρετανικός λαός και η Βρετανική κυβέρνηση θα συνεργαστούμε για να έχουμε νέες εμπορικές συμφωνίες ε, σε ηρεμία και πάρα πολύ βέβαια με, και με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου θα γίνει αυτό. Η κυρία Ραφάλσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δική μου πολιτική ομάδα συντηρητική και μεταρρυθμιστές, η ΣΥΑΡ υποστηρίζει αυτή την επιστολή και όλα τα θέματα που θίγει. Εμείς πάντα ε, πάγια υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα σημαντικότερα τώρα είναι η προστασία των εργαζομένων, αλλά και κάποια πρότυπα για την εργασία. Ο κύριος Βίλομσεν από Τικού, ευχαριστώ πολύ. Ε, ποια είναι η θέση μας. Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς το σεβόμαστε. Το θέμα είναι στο μέλλον πώς θα είναι οι σχέσεις μας. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε να έχουμε μια σχέση όπου να μην χωράει μισολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτή είναι ξεκάθαρη άποψη που εκφράζει η επιστολή, άρα και την υποστηρίζουμε. And now, Mr. Pattern, please. Uh, thank you, Chair. Um, Το θέμα το οποίο είχα θέσει στην ημερήσια διάταξη είναι ότι η επιστολή μαζί με τη γνωμοδότηση λέγει ότι εμείς ε, είχαμε κατά κάποιο τρόπο κάνει τη συζήτηση ενώ δεν το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι τέτοιο, ευχαριστώ για την πρότασή σας, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει η επιστολή δεν ε, είναι αλήθεια. Εγώ δεν μπόρεσα να συνεισφέρω στην επιστολή αυτή γιατί η διαδικασία με εμπόδισε να το κάνω. Νομίζω ότι εδώ έχει υπάρξει ένα σαφές δημοκρατικό έλλειμμα. Τώρα, ε, για την γνωμοδότηση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία με τα οποία σύμφωνο. Υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία διαφωνώ. Διαφωνώ ριζικά και διαφωνώ και με τον προηγούμενο συνάδελφο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας ε, στην ουσία ε, ξεπερνάει τις αρμοδιότητες της σχολιάζοντας τη Συμφωνία Αποχώρησης και η Επιτροπή, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή μας προσπαθεί ουσιαστικά και κάνει προτάσεις να επιβάλλει κάποιους κανόνες και νόμους σε μια χώρα η οποία θα έχει αποχωρήσει και δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Όπως είπα, εμείς έχουμε υψηλά επίπεδα προστασίας, κοινωνικής προστασίας, ελαχίστου μισθού κτλ και δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιες προσπάθειες επιβολής. Εγώ λοιπόν δεν θα υποστηρίξω την γνωμοδότηση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Πάτεν. Κοιτάξτε, εγώ δεν κανόνισα την, τους κανόνες για τη συζήτηση. Οι συνάδελφοι είπαν αυτά τα οποία θέλοντας θέλησαν να πούν. Ε, και επειδή εσείς διαφωνείτε με το περιεχόμενο της επιστολής, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν δημοκρατική η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Είναι η διαδικασία την οποία παρέχει το άρθρο 56. Δεν υπάρχει άλλη, από, αν θέλετε, υποχρέωση από πλευρά μας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν που σταθήκατε επικοδομητικά. Θα ξεκινήσουμε τώρα τις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με ηλεκτρονικές κλήσεις. Πρώτο είναι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ηλεκτρονική κλίση λοιπόν. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Ευχαριστώ. Προχωράμε τώρα στην επιστολή με την γνωμοδότηση, στην επιστολή εν πάση σχετικά με το Brexit. Ηλεκτρονική ψήφος και ονομαστική ε, επίσης ε, ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα στη ψηφοφορίας. Δεκτή. Το σημείο 10 είναι η απαλλαγή, μια πρώτη απαλλαγή για το Eurofound. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη η τροπολογία 1. Ψηφίζουμε τώρα στην συμβιβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε στην συμβιβαστική Β. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική δ. αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική C αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα τώρα της τροπολογίας 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική ή αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 και 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Τελική ψήφος τώρα, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Δεκτή. Το σημείο 11 τώρα. Απαλλαγή του Οργανισμού για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική α αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 9 λέει η πρόεδρος, όχι λάθος, διορθώνει. Συμβιβαστική β κεφαλαίο ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 6 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτή. Συμβιβαστική 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές απερίφθη D υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 18 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 και 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρας. Δεκτή. Σημείο 12. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευρωπαϊκό Δρυμαϊκό Δεσμό, συγχωρείτε. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16-17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ονομαστική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία πέρας δεκτή 13 σημείο στη μερίσια διάταξη τροπολογία 1, 1, 1, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή και ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας Δεκτεί. σημείο 14 τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ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 εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική, όχι συμβαστική, κανονική τροπολογία 25. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές ε, έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση το πρώτο μέρος της τροπολογίας 25 αρχίζει τώρα πέρασα απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με ονομαστική κλίση τώρα το σύνολο, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Περάς. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο, 15. Ορίστε. Ότι έγινε, δεν δούλεψε ο μηχάνημά σας. Ωραία. Can we repeat the vote? Μπορούμε να επαναλάβουμε την τελική ψηφοφορία. Ωραία. Αρχίζει. Και λίγη τώρα. Α, ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ωραία. Εγκρίνεται. Το 15 τώρα. Η τροπολογία 1. Ψήφι περ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική ε, Β υπέρ κατά αποχές Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 και 22 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ονομαστική κλίση για το σύνολο αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Θαυμάσια και σπουδαία. And Sorry, but we have to now get back. Λοιπόν, έχουμε και το σημείο 2. Yeah, thanks. Uh, the chair announcement. Έχουμε τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχουμε, όπως είδατε, και στις 22 γλώσσες μας διερμηνία. Έχουμε ανακοίνωση για τον οικονομικό διάλογο Apple για την ετήσια βιώσιμη ε, ανάπτυξη με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης και τους ε, ε, επιτρόπους Τζεντιλόνι και Σμιτ θα γίνει τη Δευτέρα 27 του μηνός από τις 4 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 5.30. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει μόνο η Επιτροπή ΕΚΟΝ για τα δημοσιονομικά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις 5.30 ε, μέχρι τις 6.30. Έχετε ενημερωθεί όλοι για αυτή την ε, συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τρίτον, ε, τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεών μας το Φεβρουάριο. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 18-19 Φεβρουαρίου 2020 και μας ζήτησαν να ματαιώσουμε τις συνεδριάσεις που είχαμε σε δύο μισές μέρες, στις 19 του μηνός. Ε, στις 20 δεν αλλάζει τίποτα, παραμένει η συνεδρίασή μας. Ε, ε, θα μπορούσαν να μας δώσουν, αν χρειαστούμε επιπλέον, ε, χρόνο στις 17 το μηνό το απόγευμα χρειάζεται να συνεδριάσουμε. Άρα, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου το απόγευμα η συνεδρίασή μας, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και, ε, ε, συγγνώμη, 5 και 4 το απόγευμα με 7 το βράδυ είναι το ωράριο και την 5η 20 Φεβρουαρίου πρωί και απόγευμα. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Δεν ξέρω αν έχετε προτάσεις, σχόλια κτλ. Θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Επόμενο θέμα. 5. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βάση του άρθρου 74 θα ακούσουμε πρώτα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ κύριος Κάζα είναι μας. Παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος. Όπως ξέρετε, η έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνολοκληρώθηκε στην προηγούμενη θητεία. Η διαπραγματευτική εντολή επιβεβαιώθηκε από την ψηφοφορία της Επιτροπής μας σε αυτή τη θητεία 2 Οκτωβρίου 2019 πριν από τα Χριστούγεννα ξεκίνησε ο τριμερής διάλογος και στην πρώτη συνάντηση οι συνομοθέτες καθόρισαν τις προτεραιότητες. Επίσης, δώσαμε εντολή στις τεχνικές ομάδες να ξεκινούν να αναζητούν πιθανές λύσεις ε, που θα εγκριθούν μετά σε πολιτικό επίπεδο. Ξεκαθάρισα, όπως ε, ε, είπαμε πριν, ότι είμαστε κατά της συμπερίληψης σημαντικών στοιχείων του ε, στο στο ΠΔΠ, στο διαπραγματευτικό κουτί. Θα συνεχίσουμε να συνεννόμαστε με τους ηγητές Επιτροπής Προϋπολογισμού έτσι ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Η πρώτη τεχνητή συνάντηση έγινε την προηγούμενη Δευτέρα και πρέπει να πω ότι η διαπραγματευτική μας ομάδα κάνει εξαιρετική δουλειά και σημειώνει σημαντική πρόοδο. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πληροφορίες αυτές κύριε Κάζα. Και τώρα θα ακούσουμε την κυρία Μάξοβα για την απόσπαση οδηγών. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συνοψίσω τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το πακέτο της κινητικότητας, ιδιότερα για την απόσπαση οδηγών. Το Δεκέμβριο του 19 έγινε ο τρίτος τριμερής διάλογος. Στις 11 το μηνός ήταν πολύ μακρές οι διαπραγματεύσεις και τελικά συμφωνήσαμε στα εξής. Εναρμόνιση των κανόνων των διεθνών οδικών μεταφορών, βγάλαμε από την απόσπαση τους οδηγούς φορτηγών, τα καταφέραμε. Επίσης λάβαμε υπόψη κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με ενδοομιλικές συναλλαγές. Επίσης ρυθμίζεται το θέμα των οδηγών που είναι των χωρών και ε, έχει πάει το θέμα, έχει πάρει το δρόμο του προς τη δεύτερη ανάγνωση. Και θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία και τους συνεργάτες. Φεύγει από μας το θέμα, δεν θα συμμετέχει πια η Επιτροπή ΕΜΠΛ. Στις 21 του μηνός ψήφισε η Επιτροπή Μεταφορών 27 ψήφι υπέρ 22 κατά, επί 49 παρόντων. Στις 21 Απριλίου ε, προβλέπεται νέα ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραν. Στην Ολομέλεια αναμένεται να έρθει το θέμα το Μάιο και το αργότερο τον Ιούνιο κάτι έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να πούμε ότι η θέση του Συμβουλίου ε, είναι πολύ κοντά σε εκείνη του Κοινοβουλίου για τα σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ και για τη συντομία σας. Ο κύριος Βίλομσεν, θέλετε να πείτε κάτι για αυτό το θέμα. Yes, just uh, very shortly, I would like... Πάρα πολύ σύντομα. Ε, εξ ονόματος της ε, ομάδας Ενωτικής Αριστεράς, ε, καλωσορίζουμε τις εξέλιξεις για την απόσπαση εργαζομένων, αλλά δεν θα θέλαμε να υπάρχουν παρεκκλήσεις και εξαιρέσει από τον κανόνα. Ε, αναγνωρίζουμε τη δουλειά που έχει γίνει, που ήταν πολύ σκληρές και ε, μακροσκελής οι διαπραγματεύσεις. Από όλες τις πλευρές καταβλήθηκαν προσπάθειες για να καταλήξουμε σε αυτή τη δέσμη και είναι κρίμα που ο κύριος Δομπρόφσκης, που μόλις ανέλαβε εκτελεστικός αντιπρόεδρος, προσπαθεί, ακόμα δεν ανέλαβε, να υπονομεύσει τη συμφωνία που έχουν κάνει οι συνομοθέτες. Η πράσινη ειδή και η μετάβαση και τα λοιπά. Για να είμαι ειλικρινής, αυτά είναι ανοησίες και τίποτα άλλο. Αν θέλουν κάποιες εταιρείε ε, να κάνουν καμποτάζ 8 εβδομάδες και να αλωνίζουν πάνω κάτω στα κράτη-μέλη, μπορούν να συστήσουν εκεί εταιρείε χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα του κυρίου Ντομπρόφσκη, τι έχει σχέση να κάνει με την ε, πράσινη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν μπορεί να συμβαδίζει η πράσινη μετάβαση με κάποιες εικονικές εταιρείες ε, και διάφορες παρανομίες που γίνονται. Εμείς διαφωνούμε απολύτως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Ο κύριος Ράτκε για τις ελάχιστες απαιτήσει για το μέγιστο χρόνο οδήγησης ε, των ε, και των ημερήσεων. Μπορώ να τα πω έτσι γρήγορα στα γερμανικά. Μετά από ώρες ε, διαπραγματεύσεις είχαμε κουραστεί τόσο ώστε τελικά συμφωνήσαμε και βεβαίως ο καλός συμβασμός σημαίνει ότι κανείς ε, δεν είναι εντελώς ικανοποιημένο. οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε, όλοι θα θέλαμε περισσότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα θετικό για εμάς. Ε, για εμάς ήταν σημαντικό επίσης να έχουμε ένα πλαίσιο αναφορά ε, δύο εβδομάδων, το οποίο δεν θα έπρεπε να αλλάξει και μετά από δύο εβδομάδες να υπάρξει ένα κανονικό διάλειμμα και θα δοθεί τώρα μετά από πίεση του Συμβουλίου μια εξαίρεση να υπάρξουν δύο συντομότερα διαλύματα αλλά αυτό μόνο εκτός της ε, ιδιαίτερης πατρίδας του οδηγού νομίζω λογικό είναι αυτό Τώρα για την ε, εισαγωγή νέων ε, ταχογράφων στα βαρέα φορτηγά θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2025, κάτι το οποίο επίσης είναι ιδιαίτερο σημαντικό είναι ότι έχουμε αυτή τη ρυθμίση και για τα ελαφρά φορτηγά έχουμε την εισαγωγή μέχρι το 2026 πάρα πολύ σημαντικό για τους οδηγούς αυτών των φορτηγών γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μία τάση ότι ε, βασίζονται όλο και περισσότερο στα ελαφρά φορτηγά ακριβώς για να αποφύγουν τους ταχογράφους και όλα αυτά βεβαίως τα πληρώνουν οι οδηγοί οπότε η ρύθμιση τώρα επιβάλλεται και εκεί όσον αφορά την απαγόρευση ύπνου στην καμπίνα, στα διαλύματα κτλ. Παρόλο την κριτική λοιπόν που μπορεί να ασκήσει κανείς νομίζω ότι έχουμε έναν ισορροπημένο συμβασμό. Ναι, πράγματι αυτό έχει σημασία στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περνάμε τώρα στο σημείο 16 παρουσίαση Eurovan για τα μοντέλα συλλογικών διαπραγματεύσεων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και με συγχωρείτε. Ε, ο χρόνος πιέζει. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είπατε ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Είχαμε μία μακρά παρουσίαση, αλλά θα περάσουμε γρήγορα κάποιες από τις διαφάνειες έτσι ώστε να υπάρξει και χρόνος για συζήτηση. Αυτό είναι θα έλεγα χοντρικά το πρόγραμμα το οποίο έχουμε σε σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε εξετάσει τις τελευταίες μελέτες, τις οποίες έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι, έχουμε συγκρίνει τα δεδομένα, έχουμε εξετάσει τα συστήματα των συνδικαλιστικών σχέσεων, με βάση όχι μόνο τις δικές μας μελέτες αλλά και με βάση ε, τις εργασίες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κτλ. Τώρα για να περάσω σε θέματα ουσίας. Εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα περίπλοκο, το οποίο είναι ένα σύνολο των μοντέλων ε, συνδικαλιστικών σχέσεων ή σχέσεων αντιπροσώπευσης εργαζομένων. Ε, τα εισερχόμενα είναι το γενικό περιβάλλον, οι εμπλεκόμενοι, οι διαδικασίες και για όλα αυτά οι διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές είναι πολύ σημαντικές. Και, υπάρχει και ε, τα, υπάρχουν και τα εξερχόμενα, δηλαδή τα αποτελέσματα στα εισοδήματα, στις τελικές, διαπραγματεύσεις, τελικές συμφωνίες, συμβάσεις και στην νομοθεσία την εργασιακή είναι κάτι το κεντρικό θα έλεγα για όλα τα τμήματα του συστήματος η συλλογική διαπραγμάτευση. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και τον ρόλο της νομοθεσίας και τον ρόλο της ε, διαπραγμάτευσης. Πρωταγωνιστές είναι φυσικά οι οργανώσεις των εργαζομένων, είναι οι οργανώσεις των εργοδοτών, η αυτονομία τους, η διαπραγματευτική τους δυνότητα το τομέα της διαδικασίας φυσικά είναι μια από τις πιο σημαντικές ε, η συλλογική διαπραγμάτευση. Θα έλθουμε αργότερα στα διαφορετικά επίπεδα και σε ποιο βαθμό μεταξύ τους αλληλοεπηρεάζονται. Τι ρόλο μπορεί να παίξει το κράτος, ε, ε, ας πούμε δεχόμενο αποτελέσματα διαπραγμάτευσης για μη διακανονισμένα τμήματα του χώρου της εργασίας ή δεχόμενοι τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης και για τον καθορισμό συγγνώμη, των αμοιβών. Έχουμε επίσης ε, στο τέλος και τα αποτελέσματα, δηλαδή ε, τις συλλογικές συμβάσεις και ε, την νομοθεσία την εργασιακή. Βλέπετε λοιπόν τα αποτελέσματα. Τώρα θα περάσω πολύ γρήγορα στις επόμενες δύο διαφάνειες κάνοντας ορισμένες ε, παρατηρήσεις. Βλέπουμε την πυκνότητα εδώ, ε, δηλαδή το ποσοστό των εργαζομένων που ανήκουν σε συνδικάτα. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα. Ίσως χρειάζεστε κι άλλα για να διαβάσετε βέβαια τη διαφάνεια αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι έχουμε στις βόρειες χώρες και το Βέλγιο υψηλότατα επίπεδα συμμετοχής. Ε, πολλές φορές τα συστήματα αυτά συνδέονται και με το σύστημα ασφάλισης των εργαζομένων. Υπάρχουν πολύ ε, χαμηλότερα ποσοστά στη Νότια Ευρώπη αλλά υπάρχουν και χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία που είναι σχετικά χαμηλά. Τώρα εδώ βλέπουμε τις αλλαγές στην πυκνότητα των εργαζομένων σε μία 16 ετή περίοδο. Ο κανόνας είναι γενικά πτωτικός. βλέπουμε τις κεντρικές και ανατολικές χώρες, εκεί έχουν υπάρξει σημαντικότατες μειώσεις συμμετοχής, υπάρχουν συμμετοχές μειωμένες και στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά εκεί είναι πάντα ψηλά τα ποσοστά. Τώρα, σχετικά με τις εργοδοτικές οργανώσεις, εδώ έχουμε στοιχεία από διαφορετική χρονική περίοδο και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές, ε, θα έλεγα, διακυμάνσεις Βλέπουμε εδώ το ποσοστό των εργαζομένων που ε, ε, ε, εργάζονται σε επιχειρήσεις που ανήκουν στις εργοδοτικές οργανώσεις. Εδώ βλέπουμε διαφορές ανάμεσα στην Ισπανία και την Γαλλία που έχουν χαμηλή συνδικαλιστική συμμετοχή πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Εδώ υπάρχουν επίσης ε, και κάποιες ρυθμίσεις στην Αυστρία, ας πούμε, που δίνουν αποτελέσματα 100% ε, γιατί είναι υποχρεωτικό οι επιχειρήσεις να ανήκουν στις εργοδοτικές οργανώσεις. Βλέπουμε επίσης τις χώρες οι οποίες έχουν την υψηλότερη πυκνότητα με σταθερή παραμονή στο συγκεκριμένο επίπεδο. Και υπάρχουν κάποιες ε, ποικίλε διαφοροποιήσεις. Ε, βλέπουμε ότι η, η πυκνότητα συμμετοχής στις εργοδοτικές είναι ε, μερικές φορές διαφορετική από την αντίστοιχη στις ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες και σε αυτή την διαφάνεια, τις οποίες δεν θα σταθώ. Τα μικρά τρίγωνα που βλέπετε Όσο πιο ψηλά είναι, αυτό σημαίνει ότι τόσο πιο συγκεντρωτικό είναι ε, το σύστημα των διαπραγματεύσεων στις συγκεκριμένες χώρες. Και το χαμηλότερο είναι, θα έλεγα, σε επίπεδο επιχείρησης ουσιαστικά. Βλέπουμε κάποιο συσχετισμό ανάμεσα στα επίπεδα διαπραγμάτευσης στις διάφορες χώρες Τα υψηλά επίπεδα διαπραγμάτευσης μπορεί να σημαίνουν και ε, υψηλά επίπεδα πυκνότητας των ε, πρωταγωνιστών που προείπα, αλλά μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζουν και το ρόλο του κράτους που υποστηρίζει την διαπραγμάτευση. Στη Γαλλία, σαν παράδειγμα, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, με υψηλή κάλυψη συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ το επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων στα συνδικάτα είναι χαμηλό. Ας περάσουμε γρήγορα από ορισμένε διαφάνειες, δεν έχουμε χρόνο. Τα βασικά μηνύματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε εμείς εδώ είναι ότι ενώ υπάρχει πίεση ε, σε ορισμένες χώρες, παρόλα αυτά παραμένει υψηλό σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο ε, η Γαλλία, η Πορτογαλία κτλ. Το σύστημα υφίσταται πιέσεις, αλλά οι πιέσεις αυτές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπερβολές. Ε, για τα επόμενα δύο, ε, τους επόμενους δύο πίνακες θα έλεγα έχουμε μια σχηματική διαπραγμάτευση των διαπραγματεύσεων των, σε διμερές ή τριμερές επίπεδο εδώ έχουμε κάποια στοιχεία και από την παλαιά Ευρώπη των 15. Οι συγκεντρωτικές, ε, ε, θα έλεγα, συλλογικές διαπραγματεύσεις ε, είναι οι πιο καθοριστικές. Όταν περνάμε στην επόμενη διαφάνεια, στα 13 κράτη-μέλη που ήρθαν πιο πρόσφατα στην Ένωση, το σημαντικό επίπεδο που γίνεται η διαπραγμάτευση είναι το επίπεδο της επιχείρησης. Λοιπόν, τα τελευταία λεπτά πριν δώσω το λόγο στον Christian, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες ε, τυπολογίες και κάποιες ομαδοποιήσεις χωρών. Ε, εδώ το έχει κάνει ένας γνωστός ε, επιστήμον και είναι μια δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008. Βλέπετε τις χώρες οι οποίες έχουν συνδυάσει τις προσπάθειές τους Ε, πάνε κάπως γρήγορα οι διαφάνειες. Στις βόρειες χώρες υπάρχει θα έλεγα οργανωμένο συνεταιριστικό κίνημα, ισχυρές ε, επίσης παρεμβάσεις συγκεντρωτικές ε, των εργοδοτικών εργανώσεων στην κεντρική Ευρώπη ε, το πρότυπο των κοινωνικών εταίρων χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, ασθενή συνδικάτα και ισχυρότερη εργοδοτική συσπήρωση. Ε, στο Νότο, στις περισσότερες χώρες, οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο κρατικό, ε, το φιλελεύθερο βορειοδυτικό αν θέλετε μοντέλο βασίζεται σε εθελοντικές αν θέλετε συμμετοχές, εμπλέκει εν πολύ στους κοινωνικούς εταίρους. Στην Ανατολική Ευρώπη, και αυτή είναι δουλειά του 2008 επαναλαμβάνω, έχουμε ένα συνδυασμό του φιλελεύθερου μοντέλου με το μοντέλο όπου το κράτος παίζει σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, ε, το ε, κεντρικό μοντέλο διαπραγμάτευσης στις βόρειες χώρες βασίζεται ε, στην συνεταιριστική αντίληψη για τη συμμετοχή στις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ στο κέντρο της Ευρώπης και στην Ανατολική Ευρώπη βασίζεται σε διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχείρησης. Ε, το κράτος στον βορρά έχει μειωμένη συμμετοχή αν θέλετε, ενώ στον νότο είναι συστηματική η παρέμβαση του κράτους, το οποίο παρεμβαίνει πολύ πιο συχνά ε, στις ε, κεντρικές χώρες της Ευρώπης και τις ανατολικές χώρες υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ε, θα έλεγα ότι έχουμε φιλελεύθερα πρότυπα περισσότερο στο βορρά και στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ στο νότο έχουμε πρότυπα συγκεντρωτικού τύπου ε, στις περισσότερες μορφές διαπραγματεύσεων. Τώρα για το είδο, το ύφος, ε, τη μορφή των διαπραγματεύσεων. Έχουμε σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων και σε επίπεδο συνεταιριστικό διαφορές από ό,τι έχουμε στο νότο ε, και στη Δυτική Ευρώπη. Η διαπραγμάτευση δεν έχει μόνο ε, στόχο την κατανομή αλλά και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας και αυτό συνδέεται και με την ισχυρή συμμετοχή και συσπήρωση των εργοδοτικών οργανώσεων. Τώρα, ο Κρίστιαν θα μας μιλήσει για το τι συνέβη μετά το 2008. Θα συνεχίσω λοιπόν. Ο Ντέιβιντ ανέφερε τις βασικές ε, τάσεις ε, που υπάρχουν ε, που ίσως επιταχύνθηκαν με την κρίση. Είδαμε τα τελευταία 15-20 χρόνια πρώτα απ' όλα δύο πράγματα. Την αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων από το εθνικό στο κλαδικό επίπεδο σε επίπεδο Εταιρεία. η πρώτη τάση αυτή και η δεύτερη τάση είναι η εξασθένηση των ε, συνδικάτων, δηλαδή έχει μειωθεί η συμμετοχή και πάλι επιταχύνθηκε από την κρίση και μάλλον έτσι θα παραμείνει. Δεν έχουμε δει το ίδιο πράγμα στους εργοδότες. Μπορεί να είδατε ε, το διάγραμμα πριν. Έχει μείνει σταθερή η συμμετοχή τους Δεν έχουμε λοιπόν κάποια σχετικά στοιχεία. Καθώς λοιπόν έχουν πέσει και οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις και οι συμμετοχή στα συνδικάτα έχουν παρέμβει τα κράτη σε πολλά κράτη-μέλη και βλέπουμε κάποια κρατική μονομέρεια. Ο Ντέιβιτ σας έδειξε εκεί πέρα την αύξηση από το 2008. Θεωρούσαμε ότι έπρεπε το Eurofund λοιπόν να παρέμβει και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία με νέα δεδομένα και σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Εντάξει, μοιάζει απλό τώρα αυτό που είναι στην οθόνη, αλλά το να μπορέσουμε να το απεικονίσουμε θεωρητικά ως ένα τρίποδο το οποίο προσπαθεί να εξορροπήσει τα συμφέροντα δεν είναι απλό. Στο κέντρο ε, λοιπόν ε, βλέπετε εδώ πέρα ε, την έκφραση. Λοιπόν, όλα αυτά βασίζονται σε ένα βασικό βιβλίο του κυρίου Μπάντ, Αμερικανού, Απασχόληση με ανθρώπινο πρόσωπο λέγεται και λέει ότι κάθε σύστημα εργασιακών σχέσεων θα πρέπει να εξορροπεί τρία πράγματα. Την αποτελεσματικότητα, την ισότητα και την εκπροσώπηση. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα την εκπροσώπηση, την εργασιακή δημοκρατία που βασίζεται ίσως στο παλαιότερο σχετικό ε, βιβλίο των Web, Beatrice και Sydney Web ε, που αφορούσε την εργασιακή δημοκρατία και τα συνδικάτα και μετά έχουμε τα τρία αποτελέσματα. Κοινωνική δικαιοσύνη, ποιότητα εργασίας που είναι ε, το βασικό αυτό το οποίο κάνουμε και βεβαίως ε, για τους εργοδότες, αλλά όχι μόνο για αυτούς, ε, την βιομηχανική αποτελεσματικότητα. Οπότε, το επόμενό μας ερώτημα είναι πώς θα τα μετρήσουμε αυτά. Ήμασταν κάπως επιφυλακτικοί στην αρχή, αλλά με τη βοήθεια διακεκριμένων ε, ακαδημαϊκών ε, μιας ομάδας Ισπανών καταλήξαμε σε έναν δίκτυ εργασιακών σχέσεων ε, τώρα και πάλι δεν μπορείτε να το διαβάσετε ίσως είναι πολύ μικρό καταλήξαμε σε 13 δίκτες εργασιακής δημοκρατίας δηλαδή συμμετοχή στα συνδικάτα, κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις μετά έχουμε ένα μέσο επίπεδο και μετά έχουμε το επίπεδο της εταιρείας ε, που βασίζεται κυρίως στις έρευνές μας, πληροφορίες που δίνεται στα συνδικάτα, συμβούλια εταιρικά και έτσι έχουμε φτιάξει έναν δίκτυ τον οποίον λέμε δίκτυ εργασιακής δημοκρατίας. Έτσι καταφέραμε μετά να έχουμε μεγαλύτερες λεπτομέρειες ε, ε, κάποια από αυτά παρέμειναν ίδια, κάποια είναι πιο ενδιαφέροντα. Έχουμε λοιπόν έξι δέσμες. Ε, το ένα είναι κοινωνική εταίρη, δεύτερη κορπορατισμός, ε, τρίτον μια διοίκηση σε ένα κρατικό πλαίσιο. Το 4 και το 5 θα είναι κάποια μοντέλα που βασίζονται στην εταιρεία, είτε στο καταστατικό της εταιρεία είτε πιο εθελοντικά. Και το έκτο είναι κάτι το οποίο είναι προσανατολισμένο στην αγορά και με βάση αυτά μπορέσαμε να δούμε το πόσο αποδίδουν τα μοντέλα αυτά. Έχουμε λοιπόν την μετακίνηση της Γερμανίας από το κοινωνικό μοντέλο στο εταιρικό μοντέλο και μπορέσαμε επίσης να δούμε κάτι το οποίο δεν είχε κάνει ο Βίσερ τα νέα κράτη-μέλη τα οποία ο Βίσερ είχε βάλει σε ένα τσουβάλι ήταν κάπως χοντρικό αυτό βλέπετε τώρα ότι ε, εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία. Παραδείγματο χάρη στο 4 βλέπετε Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβακία. Ναι, εντάξει. Βλέπουμε μετά στο 6 όπου υπάρχει ένας προσανατολισμός στην αγορά προφανώς στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η Εστονία και η Πολωνία που έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Οπότε τι έχουμε μετά εδώ πέρα, τους κοινωνικούς εταίρους, ε, την κλασική περίπτωση, υψηλό βαθμός ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων, ε, με συγκεντρωτική δομή, τα πάνε καλύτερα στην εργασιακή δημοκρατία ε, Βεβαίω είναι ακόμη ασθενή τα συνδικάτα, πολύ ισχυροί οι εργοδότες, 100% ε, κάλυψη από συλλογικέ διαπραγματεύσεις, επειδή υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή των ε, επιχειρήσεων, του χάρη στο Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο. Πώς πάει η κατάταξη λοιπόν, το μπλε είναι ο μέσο όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κόκκινο είναι η περίπτωση αυτή που είπαμε, οι κοινωνικοί εταίροι. Τα πάνε καλύτερα σε όλες τις διαστάσεις. Το άλλο είναι κορπορατισμός. Μοιάζει με το προηγούμενο σύστημα. Υπάρχει μεγάλος σχετισμός μεταξύ λογικής αυτονομίας και κοινωνικών εταίρων. Οπότε, εδώ μιλάμε κυρίως για τις σκανδιναβικέ χώρες, ε, πολύ κοντά στο προηγούμενο μοντέλο, αλλά οι κοινωνικοί εταίροι είναι πιο αυτόνομοι Έχουμε λοιπόν συμβούλια εργαζομένων ισχυρά με δικαίωμα συναπόφαση σε επίπεδο εταιρεία και αυτοί τα πάνε καλύτερα όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο. Τώρα το πώς θα πάνε ε, και πάλι μπλε είναι ο μέσος όρος, το κόκκινο είναι το συγκεκριμένο μοντέλο Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Σουηδία ε, πάνω από τον μέσο όρο. Το τρίτο είναι, με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος, αν έχετε την καλοσύνη να μιλάτε λίγο πιο σιγά για να σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Έχουμε μια διοίκηση σε ένα κρατικό πλαίσιο. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ο ρόλος που παίζει το κράτος εδώ χαμηλή συμμετοχή στα συνδικάτα, αλλά τα πηγαίνουν αρκετά καλά οι εταιρείε. Μάλλον χαμηλά είναι η απόδοση του κοινωνικού διαλόγου παρά το ότι υπάρχουν εταιρικά συμβούλια. Δηλαδή θα λέγαμε Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα και έχουμε ισχυρό ρόλο του κράτους και πώς θα πάνε ε, βρίσκονται γύρω στον κοινοτικό μέσο όρο. Και τέλος Εστονία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, ε, προσανατολισμένες στην αγορά, λιγότερος ε, ρόλος ε, των κοινωνικών εταίρων, μικρότερος και εργοδοτών και εργαζομένων έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία εργασιακής δημοκρατίας και εδώ βλέπετε πως τα πάνε ε, λοιπόν, ε, μιλάμε για συσχέτιση. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει αιτιώδης ε, σχέση και κατά κάποιον τρόπο αποδίδει εξίσου καλά το μοντέλο με χαμηλότερη εργασιακή δημοκρατία. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς αυτά τα πράγματα. λοιπόν, εξετάσαμε κάποια φαινόμενα με βάση τα δεδομένα. Τα εξετάσαμε σε κάποια χρονική στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αιτιώδη σχέση. Οπότε το πλαίσιο αυτό είναι αυτό το οποίο είναι με τα υπέρ και τα κατά του. Έχουμε επιτύχει όμως δύο πράγματα για πρώτη φορά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας δείκτης εργασιακών σχέσεων και δεύτερον ε, μπορούμε να τα δούμε αυτά πιο λεπτόμερως με βάση τα δεδομένα μας. Μετά, μια που μιλάμε για συσχετισμούς, όταν διασταυρώνουμε τα δεδομένα αυτά με, άλλα, με άλλους δείκτες, βλέπουμε δύο πράγματα ότι οι χώρες οι οποίες έχουν τον υψηλότερο βαθμό εργασιακής δημοκρατίας είναι αυτές με την υψηλότερη βαθμολογία στην αποτελεσματικότητα. Και το δεύτερο, ε, το είπε ήδη ο Ντέιβιντ, φαίνεται ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του επίπεδου συλλογικών διαπραγματεύσεων και της απόδοσης. Δηλαδή, οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλότερο επίπεδο συλλογικών διαπραγματεύσεων ε, φαίνεται ότι τα πηγαίνουν καλύτερα στο επίπεδο της εργασιακής δημοκρατίας. Αλλά όπως σας είπα, είναι συσχετισμός και όχι αιτιώδης σχέση. Αυτά. Ελπίζω να ψάμε και ώρα για συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε και πλούσια σε στοιχεία. Ερωτήσεις από τα μέλη. Κύριος Πισλάρου, πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ χρήσιμα αυτά, γιατί είναι πολύ σχετικά με τα θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του έτους. Κατώτατος μισθός και άλλα uh, για την ε, ε, εργασιακή δημοκρατία. Έχουμε άλλα δύο μοντέλα, αλλά δεν είδαμε τις γραφικές ε, παραστάσεις. Υπάρχει καμία εξήγηση, ήταν τόσο χάλια που δεν βλέπονται και δεν μπορούσατε να τα ε, παραστήσετε γραφικά, μπορείτε να μας τα στείλετε με σχόλια για να έχουμε το πλήρη ε, κατάλογο και να μπορέσουμε να συγκρίνουμε. Και κάτι άλλο που βοηθήσατε ότι πρέπει να κάνουμε εμείς οι πολιτικοί. Δεν βλέπω συστάσεις εδώ για πολιτική. Ε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ε, τι έχετε μελετήσει, πού έχετε καταλήξει. Ξέρω ότι αν είχατε περισσότερο χρόνο θα τα λέγατε αυτά. Ε, αυτή η εργασιακή δημοκρατία είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να αγωνιστούμε. Είπατε ότι υπάρχουν χώρες που αποδίδουν χωρίς να είναι στο καλύτερο μοντέλο. Εσείς τι έχετε να προτείνετε και όλα αυτά. Ε, ε, πρώτα θα συλλέξουμε τις ερωτήσεις και μετά θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε. παρακαλώ. Ε, ο κύριος ε, Άγγελ, ε, Ευχαριστώ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, λέει ο κύριος Άγγελ, να μαθαίνουμε τι λέτε. Ε, αναφερθήκατε σε αυτές τις εξενότητες, τα κλάστερ, και η Γερμανία έχει αλλάξει κατηγορία από τη σχέση κοινωνικών εταίρων στον οργανωμένο κορπορατισμό. Τώρα, αυτή η χώρα έχει μια πολιτική σταθερότητα. Για ποιο λόγο άλλαξε μοντέλο. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν γνωρίσει άλλες αλλαγές και αλλού αναμένονται ε, μετατοπίσεις. Ε, μία εξήγηση μπορεί να είναι η αλλαγή πολιτικής σε μια χώρα. Δηλαδή όταν αλλάζει η πολιτική πλειοψηφία, αλλάζει και το μοντέλο, το κοινωνικό και αλλάζει και κλάστερ η χώρα. Η κυρία Πίτερ Χάνσεν, ευχαριστώ πολύ. Ε, μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο ακριβώς η Γερμανία έχει αλλάξει κατηγορία. Και επίσης, Δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει και στις έρευνες σας. Τι γίνεται με τα επίπεδα των μισθών και τα επίπεδα των τιμών. Έχει σχέση αυτό με το ε, σε ποια κατηγορία κατατάσσονται οι χώρες. Η κυρία Περέρα, ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Εγώ είμαι από την Πορτογαλία. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές στη χώρα μου διότι ενθαρρύνουν τη συμμετοχική δημοκρατία και είναι και ένας ε, τρόπος να ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις. Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων που είναι ε, προϊόν σκληρών αγώνων. Οι συλλογικές συμβάσεις καταπολεμούν την επισφάλεια στην εργασία και εδώ βλέπουμε ένα συσχετισμό ανάμεσα στην αύξηση της επισφάλειας και τη μείωση, ε, την υποχώρηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες και οι νέοι είναι πολύ εκτεθειμένοι στην ε, επισφάλεια. Οι συλλογικέ συμβάσεις δεν θα ήταν εγγύηση προστασίας των εργαζομένων από τέτοιες ε, εξαιρετικά επισφαλείς εξέλιξη. Κυρία Φράνσεν, ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα και πρόσφατα στον κοινωνικό οδικό χάρτη που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα προτείνει μέτρα για ε, να επεκταθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και να καλύπτουν τους εργαζομένους επιγραμμικές πλατφόρμες. Εσείς πώς το βλέπετε. Και δεύτερον, η ενθάρρυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ε, στην αρχή παριθμών 8 του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Μόλις 16 όμως κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση του ILO 181 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ποια είναι τα πιο ρεαλιστικά κατά την ε, γνώμη σας σενάρια για να εφαρμοστούν ε, αποφασιστικά και αποτελεσματικά αυτές οι προτάσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε ήδη μέχρι τώρα. Η πρώτη παρατήρηση ίσως να μην έχω συμφωνήσει, όχι με την εξήγηση την οποία κάνατε εσείς, αλλά αυτά που λέει ο Βίσερ σχετικά με τις νο, νότιες δημοκρατίες και τον διαβημένο ρόλο του κράτους. Ε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Στην Ιταλία δεν είναι αλήθεια ότι το κράτος έχει ένα διαβημένο ρόλο. Υπάρχει ένα μίξ θα έλεγα, ένα ανάμεικτο σύστημα για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Και το δεύτερο θέμα, διαρωτώ με αν από επιστημονικής απόψεως και όχι πολιτικά βέβαια, εξετάσει το συσχετισμό ανάμεσα στην ισχύ του συστήματος διαπραγματεύσεων συλλογικών και την δυνατότητα εισαγωγής του μέτρου του ελαχίστου μισθού. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εκεί όπου το σύστημα των διαπραγματεύσεων είναι ισχυρό και θεσμοποιημένο, είναι πιο δύσκολο θα έλεγα και αντιμετωπίζουμε περισσότερα προβλήματα για την εισαγωγή νομοθετικών μέτρων σχετικά με τον ελάχιστο μισθό. Ενώ το αντίθετο ίσως να είναι ε, πραγματικό με λοιπόν αν έχετε ε, σκεφτεί λίγο τον συσχετισμό αυτό. Η κυρία Μπρινέ και μετά η κυρία Σντάνοκα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Η ερώτησή μου ήταν αντίστοιχη με αυτήν η οποία μόλις τέθηκε σχετικά με την άποψή σας για τα συστήματα των διαπραγματεύσεων και τις μεθόδους των συλλογικών διαπραγματεύσεων ε, και το ελάχιστο ευρωπαϊκό ε, μισθό. Η κυρία Σντάνοκα. Ξέρω ότι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης το πρόβλημα των ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, ιδιαίτερα και στις χώρες των Βαλτικών κρατών. Ε, και τα διαγράμματα τα οποία θα έλεγα μας δείξατε αναφέρονται σε αυτό. Με εκπλήσει όμως ότι η Εσθονία διαφοροποιείται από τη Λετωνία και τη Λιθουανία στην τελευταία διαφάνεια. Μπορείτε να μου δώσετε κάποια εξήγηση για τη διαφοροποίηση αυτή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τις οποίες θέσατε. Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις σύντομα. Ναι, η, η άποψη του Eurofund είναι ότι ο κοινωνικός διάλογος ε, είναι θα έλεγα ε, τμήμα αναπόσπαστο της ε, παράδοσής μας, του γενετικού μας κώδικα και είναι το κατεξοχήν μέσο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε σε διαφορετικά επίπεδα ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επηρεάζουν την διακυβέρνηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των ε, σχέσεων εργασίας τους. Θα προσπαθήσω να είμαστε ειλικρινείς. Βλέπουμε το συσχετισμό ανάμεσα στην δημοκρατία στις συνδικαλιστικές σχέσεις και την αποδοτικότητα. Στην καλύτερη περίπτωση, ε, ή μάλλον στη χειρότερη περίπτωση, δεν βλάπτει, αλλά μπορεί να βοηθά και θα πρέπει να υπάρχει μια θα έλεγα α, ισορροπία, μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην αποδοτικότητα από τη μία και την δημοκρατία, την εργασιακή από την άλλη. Υπάρχουν παραδείγματα όπως η Γερμανία. Θα μπορούσαμε να δείξουμε και κάποιους επιπλέον δείκτες οι οποίοι όμως δεν είναι ακριβώς μετρήσιμοι και θα μπορούσαμε απλά ε, να μιλήσουμε για το πόσο επηρεάζουν οι απεργίες τα πράγματα. Είναι καλό, είναι κακό, αλλά αυτό το κρίνει ο καθένας διαφορετικά ανάλογα με την πολιτική του τοποθέτηση. Δεν χρησιμοποίησαμε λοιπόν την απεργία ως δείκτη. Βλέπουμε ότι η Γερμανία σε σχέση ε, με τους μηχανισμούς τους οποίους χρησιμοποιεί ε, και σε σχέση με τον ελάχιστο μισθό, ο οποίος στην Γερμανία εισήχθη θα έλεγα πάρα πολύ πρόσφατα, μοιάζει με το συνδικαλιστικό πρότυπο λοιπόν η Γερμανία. Το θέμα είναι ότι στο πλαίσιο το οποίο εμείς χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία της Γερμανίας τα εντάσσουμε σε συγκεκριμένες δέσμες οι οποίες μεταξύ τους είναι κοντά. Ε, οι επόμενες ε, δύο δέσμες ε, δεν είναι ιδιαίτερα σε κακή κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά δεν είχαμε το χρόνο να τα αναλύσουμε αυτά πιο πολύ. Τώρα, η σύνδεση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του ελάχιστου μισθού. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση που θα πρέπει να γίνει στο μέλλον Έχετε κυρίως τις σκανδιναβικές χώρες όπου υπάρχουν ισχυροί κοινωνικοί εταίροι, όπου δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός. Ε, πολλοί πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να είναι στα πλαίσια της αυτονομίας των εργαζομένων, δεν θα πρέπει να καθορίζεται εκ των άνω. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένας συσχετισμός ανάμεσα στα δύο για την παρατήρηση της Ιταλίας. Η Ιταλία είναι λίγο εξωτική θα έλεγα σε σχέση με τις δέσμες τις οποίες ε, παρουσίασα. Έχετε το κράτος που παίζει σημαντικό ρόλο, έχετε όμως και σημαντικούς ε, κοινωνικούς εταίρους και οι συμφωνίες, ε, οι συμβάσεις του 18 αποδεικνύουν πόσο ακριβώς οι κοινωνικοί εταίροι παίζουν ρόλο. Αυτά τα υπόλοιπα ο συνάδελφος. Ε, θα κάλυψες ε, ορισμένα από αυτά που ήθελα να απαντήσω εγώ. Ε, περισσότερες πληροφορίες φυσικά μπορούμε να σας δώσουμε με μεγάλη μας χαρά. Και διμερώς αν θέλετε. Και μέσω της ε, γραμματείας, αν είναι έτσι η πιο επίσημη οδός αυτή. Ε, για την ερώτηση της κυρίας Γκολμίνη που θα μπορούσαν να είχαν κάνει και άλλοι από άλλες χώρες. Αυτό είναι μια άσκηση απλούστευσης όπου χάνονται κάποιες ιδιαιτερότητες και αποχρώσεις ε, στην προσπάθεια της απλούστευσης. Είναι πολύ σωστό πάντως το σχόλιο σας. Για τα πραγματικά επίπεδα μισθών δεν έχουμε εκεί στοιχεία. Τα συστήματα διαπραγματεύσεων και τα μακροοικονομικά αποτελέσματα ε, είναι αντικείμενο μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει μια σχολή σκέψης που λέει ε, όταν οι συλλογικές συμβάσεις αποκεντρώνονται, αυτό έχει καλύτερο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα προ προς την απασχόληση. Βέβαια η απάντηση θα ήταν ε, ότι έχει καλύτερα μακροοικονομικά αποτελέσματα με το συντονισμό των συστημάτων συλλογική διαπραγμάτευση, ανεξάρτητα από το επίπεδο αμοιβών. Για του εργαζομένου ηλεκτρονικέ πλατφόρμε και τι συλλογικέ διαπραγματεύσει δεν έχω καθόλου απάντηση. Διαβάζω διάφορα στι εφημερίδε για κάποιε απόπειρε να οργανωθούν ε, και να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι εκεί με συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα και ξέρω ότι είναι και τμήμα της ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν υποσχεθεί ότι θα κάνουν μια σύνοδο κορυφής ε, για τους εργαζομένους εκεί και η Eurofound και άλλες οργανώσεις εταίροι μας έχουν ε, πολύ υλικό. Αν θέλετε να σας ενδιαφέρει μπορείτε να το βρείτε. Για τις συστάσεις. Στον κανονισμό μας στόχο έχουμε να προωθήσουμε το διάλογο ανάμεσα στην εργασία και την εργοδοσία, τη, τη δείξη επιχειρήσεων. Φυσικά έχουμε και συστάσεις να κάνουμε. Τρεις είναι οι τομείς που έχει σημασία να δώσει κανείς προσοχή. Το πρώτο είναι να βελτιώσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της διαπραγμάτευσης. Το δεύτερο είναι η ίσχυση της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και το τρίτο που συνδέεται με τα δύο προηγούμενα η δημιουργία ικανοτήτων για τον κοινωνικό διάλογο και τους κοινωνικούς εταίρους. Και αυτό σημαντικό για σας. ανακάλυψα δύο σημεία που δεν είχαμε απαντήσει, λέει ο κύριος Βέλτς. Το πρώτο ήταν για την Εσθονία. Βεβαίως, ο Γέλε Βίσερ έχει εντάξει και τις τρεις βαλτικές χώρες ε, στην ενότητα των νέων κρατών μελών. Εμείς χρησιμοποιώντας 13 δείκτες όμως, για τις εργασιακές σχέσεις και αυτό μας έδειξε ότι είχε πιο πολλά κοινά με την Πολωνία και τη ε, Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εστονία, παρά με τη Λετωνία και τη Λιθουανία. Και το πώς θα προωθήσουμε τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις που ρωτήσατε, ε, με βάση την Σύμβαση 181 του ΆΕΛΟ Δύσκολο. η οργάνωσή μας στο Eurofound συμμετέχει στις τριμερείς διαπραγματεύσεις και μπορούμε να βοηθήσουμε. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αυτονομία και την παρέμβαση, όπως υπόθηκε. Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Από τη μια θέλουμε να προωθήσουμε τις συλλογικές, διαπραγματεύσει, αλλά από την άλλη πρέπει να είναι και αυτόνομη η κοινωνική εταιρεία. το τελευταίο βήμα θα πρέπει να το κάνουν κοινωνικοί εταίροι σε όποιο επίπεδο θεωρούν είναι το καλύτερο στο εθνικό του σύστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν μιλώ μόνο για το περιεχόμενο αλλά και για την παρουσίαση, για τον τύπο. Πραγματικά ήταν ε, μια αφύπνιση, μας άνοιξε τα μάτια. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία που μας φέρατε, γιατί χρειαζόμαστε στοιχεία και δεδομένα για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Μόνο εφόσον συζητούμε βάση περιστατικών δεδομένων και στοιχείων, μπορούμε να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Είδαμε τα διάφορα πρότυπα και μοντέλα διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούν αυτά να οδηγήσουν και να βοηθήσουν στη συζήτηση. Είναι μεγάλη η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό. Δύσκολο θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο πλαισίου και μόνο θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και θα τα ξαναπούμε στο επανειδήν.